Bene, noi possiamo cominciare. Μπορούμε να αρχίσουμε διότι έχουμε μία συζήτηση και μακροσκελή και ενδιαφέρουσα. Οπότε χρήσιμο είναι να χρησιμοποιήσουμε όλο το χρόνο. Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται στο φάκελό σας και αν δεν υπάρχει αντίρρηση θα εγκριθεί. Αύριο, και σήμερα και αύριο, έχουμε αυτήν την ε, αίθουσα στη διάθεσή μας γιατί ξέρετε με το πρόβλημα που υπάρχει από το άλλο κτίριο και ανησυχώ ιδιαίτερα με ενοχλεί μάλλον ιδιαίτερα γιατί αύριο ψηφίζουμε και δεν ξέρω πώς θα ψηφίσουμε εδώ σε αυτή την αίθουσα διερμηνία έχουμε σε όλες τις γλώσσες Όσον αφορά το ΣΕΟΠ 18, Ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές έχουν προετοιμάσει ε, μία έκθεση για την Ήτρε, μια γνωμοδότηση εν ώψη της ε, Ντόχα. και θα το συζητήσουμε αύριο υπό το κεφάλαιο προφορικές ερωτήσεις. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι το ευρωπαϊκό κανάλι Άρτε ζήτησε επειδή κάνουν ένα ντοκιμαντέρ για την ενέργεια να παρακολουθήσουν τη συνεδρίασή μας αύριο το απόγευμα κατά τη συζήτηση της έκθεσης Ρόιλ θα είναι παρόντες στη συνεδρίασή μας. Μα δεν λειτουργεί αυτό, αλήθεια λέει ο πρόεδρος. Α. Φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργεί. Θα χρησιμοποιήσω το άλλο μικρόφωνο. Ξεκινάμε τώρα την κοινή συζήτηση. Και για αυτήν τη συζήτηση έχουμε τρεις ώρες στη διάθεσή μας. Μέχρι τις έξι μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα. Τελικά θα έχουμε πια την ηρεμία να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Έχουμε οργανώσει τέσσερις ενότητες για τη συζήτηση. Το, το πρώτο μπλοκ αφορά στην Τερέζα Ριέρα Μαδουρέλ. Μετά είναι η κυρία Καρβάγιο, μετά είναι ο Έλερ, μετά είναι ο Λάμπερτς, μετά είναι ο Ματίας και ο τελευταίος είναι ο Σκίνερ με 20 λεπτά στη διάθεσή του. αυτή η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων ε, για τις ε, τροπολογίες πρέπει να λάβει υπόψη τις πιο αμφιλεγόμενες τροπολογίες αλλά και τις γνωμοδοτήσεις. Επίσης οι συνάδελφοι θα πρέπει να μας πληροφορήσουν ε, για το πώς έχουν προχωρήσει με τους συμβιβασμούς και ποια είναι η κατάσταση μέσα στις συνεδριές των σαντο. Τελείωσε αυτή η εισαγωγή. Σήμερα έχουμε και δύο ομάδες επισκεπτών προσκεκλημένους της κυρίας Καρβάλιο και προσκεκλημένους της κυρίας Νίμπλερ και δίνω το λόγο για πέντε λεπτά στη συνάδελφο Ριέρα Μαδουρέλ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν αρχίσουμε να συζητάμε τις τροπολογίες, επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να τονίσω το πνεύμα συνεργασίας με το οποίο προχωρούμε στη διαπραγμάτευση των συμβιβαστικών τροπολογιών, τόσο για τη δική μου έκθεση, όσο και για τις εκθέσεις ε, των συναδέλφων όπως ας πούμε του κυρίου Έλεγ και για τους κανόνες συμμετοχής και τη συναδέλφου Καρβάλιο. Εμείς προχωρούμε ενωμένοι για να οικοδομήσουμε μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου υπέρ της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας. Κατά την τελευταία ανταλλαγή απόψεων πρέπει να σας πω με ευχαρίστηση ότι καταλήξαμε συμφωνώντας στα περισσότερα άρθρα του κανονισμού. Προχωρήσαμε επίσης για το άρθρο 16 που αφορά στις ηθικές αρχές και στο άρθρο 19 για τα PPPs στον κανονισμό για τον ορίζοντα 2020 και τους όρους συμμετοχής, τους κανόνες συμμετοχής για το θέμα της ανοιχτής πρόσβασης στις δημοσιεύσεις που χρηματοδοτούνται από τον ορίζοντα 2020 έχουμε σχεδόν φτάσει στην εξέβρεση λύσης, μια ισορροπημένη λύση που θα επιτρέψει στην Επιτροπή να διευρύνει αυτή την αρχή. Όταν μιλάμε εμείς για ανοιχτή πρόσβαση, θέλουμε να βελτιώσουμε την επιστημονική πρόοδο και την καινοτομία και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τη δημόσια δαπάνη. Θα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες τον εσωτερικό προϋπολογισμό του προγράμματος και να σας πω ποια είναι γενικώ η θέση της ομάδας μου. Εμείς πρώτα θεωρούμε ότι οι δράσεις μαρικυρί πρέπει να έχουν περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι ένα αίτημα της επιστημονικής κοινότητας και η ομάδα μου θεωρεί ότι είναι ένα σταυρικό μέσο για την ολοκλήρωση ενός ευρωπαϊκού συστήματος έρευνας και ένα σημαντικό στοιχείο για την διάδοση της αριστείας. Το ίδιο μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και για τις ευρωπαϊκές υποδομές της e-infrastructure που στην πρόταση της Κομισιόν αντιπροσωπεύονται. Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων υπάρχει μία πλειοψηφία που θέλει να αυξήσει τον προϋπολογισμό του στόχου 3 για την ενέργεια και υπάρχει μία κάποια διαφορά με τον προϋπολογισμό, την Επιτροπή Προϋπολογισμών που θέλει να επικεντρωθεί στους στόχους 6 και 7. Η ομάδα μου θέλει ευελιξία, εσωτερική ευελιξία, αλλά θεωρεί όμως ότι είναι εξίσου σημαντικό να έχουμε και την απαραίτητη σαφήνεια. Εμείς δεν μπορούμε στους κοινωνικούς στόχους να αφιερώνουμε πόσα τα οποία δεν θα ανταποκρίνονται μετά με τις προκηρύξεις. Γι' αυτό λοιπόν στο μέσο των ΜΜΕ και στα EIT θέλουμε να έχουμε κάτι το προκαθορισμένο και πιστεύω ότι έχουμε πλειοψηφία από ό,τι είδαμε από τις τροπολογίες στη δική μας θέση. Κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, εργαζόμαστε εντατικά για να έχουμε βρία συμφωνία. Διότι το Κοινοβούλιο μιζάρει πραγματικά στην έρευνα και στην καινοτομία ως μέσο εξόδου από την κρίση. Είναι απαράβατος όρος η έρευνα και η καινοτομία για να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Ένωση πρέπει να ανταγωνιστεί με ιδέες, με υπηρεσίες και προσωποποιημένες υπηρεσίες, με γνώση και η ε, επιστήμη ως παραγωγός γνώσης και η ικανότητά μας να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση στον τομέα των προϊόντων και των υπηρεσιών και να τους βελτιώσουμε για να τους εντάξουμε στην παγκοσμιοποιημένη αγορά αποτελούν πλούτο για μας. και το Συμβούλιο πρέπει να δεχθεί ότι τέτοιες δύσκολες ώρες θα πρέπει πραγματικά να στοιχηματίσει, να βασιστεί στην έρευνα και στην καινοτομία για να προχωρήσουμε σε μια οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση. Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν θα πρέπει να επηρεάζει εκείνους τους τομείς όπως η έρευνα, η παιδεία και η καινοτομία εγγυώνται την δυναμική ανάπτυξη και τον, την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό είναι το καθαρό και εξάστερο μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλει αυτό το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρβάλιο έχει το λόγο. Καλό σας απόγευμα, Πρόεδρε Σατόρη, κυρίες και κύριοι ξεκινώ ευχαριστώντας τους συναδέλφους με τους οποίους εργάστηκα πρώτα απ' όλα σε στενή συνεργασία για τον ορίζοντα 2020. Την κυρία Διέρα Μαντουρέλια και συνάδελφο θέλω να αναφέρω ξεχωριστά για το ανοιχτό πνεύμα και την προσέγγιση αυτής της συνεργασίας. Εργαζόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα αυτής της έκθεσης για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έκθεση της ε, κυρίας Ριέρα Μαντουρέλ και το θέμα του κυρίου Έλισσα ε, σε πολύ στενή συνεργασία συνεργαζόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές για την πολύ σκληρή δουλειά που έκαναν και τα επικοδομητικά σχόλια τους και όλους τους συμβούλους ε, για πολύ σημαντική βοήθεια που έδωσαν. Επίσης θα ήθελα να σας δώσω μια επισκόπηση για τις πρόοδους που επετέχθησαν σε σχέση με το σχέδιο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα για την υλοποίηση του ορίζοντα 2020 από την τελευταία μας συνεδρίαση όταν είχαμε την πρώτη εξέταση τροπολογιών. Σε σχέση με την πρόοδο που επετεύχθη λοιπόν μέχρι σήμερα, ενώ εργαζόμαστε σε συμβαστικές τροπολογίες τώρα πλέον, έχουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είχαμε πάνω από 900 τροπολογίες όπως γνωρίζετε εργάστηκα επί 27 συμβιβαστικών τροπολογιών. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να συμπεριληφθεί ό,τι γίνεται σε σχέση με αλλαγές που προτείνουν οι συνάδελφοι χωρίς να αγνοήσουμε τη σωστή επικέντρωση που πρέπει να έχει αυτή η έκθεση σε συγκεκριμένα θέματα και να μην καλύπτει επί του επιστητού θέματα. Οι δύο αυτές εκθέσεις, η δική μου και της κυρίας Τερέσα Διέρα Μαντουρέλ, αυτές οι δύο εκθέσεις συζητούνται στο ίδιο πλαίσιο, απόλυτα στο ίδιο πλαίσιο και στις τεχνικές συνεδριάσεις και σε σχέση και με τις ε, συναντήσεις των σχεδόν συντονιστών από κοινό, όταν έχουμε ευρύτερα θέματα όπως τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Πάλι έχουμε κοινέ συνεδριάσεις ε, με την ε, έκθεση και τα θέματα του κυρίου Έλλης για τους κανόνες και κανονισμού συμμετοχής. Με αυτόν τον τρόπο, όπως ανέφερε η κυρία Ριέρα Μαντουρέλ, υιοθετούμε μια ισχυρή στεναρή θέση για τις τρεις αυτές εκθέσεις ως Ευρωκοινοβούλιο. Τα περισσότερα θέματα έχουν κλείσει. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας απλά και μόνο στο ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί και εργαζόμαστε επί αυτού, επ' αυτού ακόμα. Όπως είπε η ίδια η Τερέζα για την προσπελασιμότητα, την ανοιχτή πρόσβαση και όσον αφορά και τις δημοσιεύσεις βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια τελική διατύπωση που θα δώσει την λύση όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης, ανοιχτής πρόσβασης σε δημοσιεύματα με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αηφορία και έτσι να μπορούμε από το σημερινό σύστημα να περνάμε στο ανοιχτό σύστημα δημοσίευσεων. Συνεχίζουμε τη δουλειά για τη διαδικασία των ανοιχτών ε, στοιχείων, open data. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα στις επόμενες συνεδριάσεις σε σχέση με το κείμενο και για τα research data, τα δεδομένα που αφορούν την έρευνα Συζητούμε επίσης να δούμε ποιος είναι ο το καλύτερο μέρος για να διασφαλίζεται η συμμετοχή από τους πολίτες, να διευρυνθεί η συμμετοχή αυτή από ό,τι ε, ξέρουμε σε μικρό, μικρά κέντρα μικρότερων πανεπιστημίων, μικρότερα θεσμικά όργανα και πού θα μπορούσε αυτό να γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Στον πρώτο πυλώνα, υπό τους όρους μιας ε, οριζόντιας εργαλειοθήκης, toolbox Συζητούμε να βρούμε επίσης τον καλύτερο τρόπο ώστε να συνδεθεί η επιστήμη με την κοινωνία. Στον πυλώνα 1 ίσως ή μήπως στον πυλώνα 3 στις ε, κοινωνικές ε, προκλήσεις ή στο, σε ένα οριζόντιο πάλι σε μια οριζόντια προσέγγιση εργαλειοθήκης. Θα πρέπει να δούμε και τα θέματα των κονδυλίων, προκαθορίζοντας για παράδειγμα τα ανανεώσιμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εργαζόμαστε ακόμα, δεν υπάρχουν διαφωνίες, αλλά υπάρχουν τριβές που πρέπει να επιληθούν, προβλήματα που πρέπει να επιληθούν. Και το θέμα των βλαστοκυτάρων. Υπάρχει γενικότερη συμφωνία, θα έλεγα, μεταξύ των εισηγητών και σχεδόν εισηγητών, ότι θα έπρεπε αυτή η διεργασία να ισχύει όπως στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη με την ηθική δεοντολογία όπως έχει προταθεί. Υπάρχουν όμως κάποια, κάποιες διαφορετικές απόψεις από τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές και απόψεις από την νομική επιτροπή που βαίνουν μια διαφορετική, διαφοροποιημένη κατεύθυνση. Επίσης σε σχέση με την ε, ιατρική όσο έχει σήμερα και τις παρατηρήσεις, όλα αυτά δείχνουν ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση προσπάθειες από πλευράς ε, εισηγητού και ελπίζουμε ότι αυτό το θέμα θα μπορέσει να επιληθεί και με τις γνωμοδοτήσεις των διάφορων διαφορετικών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Νομίζω έχουμε σημειώσει αρκετή σημαντική πρόοδο. Κάποια σημεία πρέπει να καλυφθούν και να ολοκληρωθούν ακόμα και να, για να κλείσουν. Αλλά υπάρχει γενικότερη συμφωνία επ' αυτών των σημείων. Το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας αφορά τον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε επαρκή προϋπολογισμό για να χρηματοδοτηθεί αυτό το πρόγραμμα, που είναι ένα καλά σχεδιασμένο και φιλόδοξο πρόγραμμα, κάτι πολύ περισσότερο από το 7ο πρόγραμμα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Καινοτομία, έρευνα, ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει πολλά μέσα στους άξονες που έχει και για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη να βοηθηθεί η Ευρώπη να αντιμετωπίσει την κρίση που διανύει. Ελπίζουμε φυσικά ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να συμφωνήσει και εκείνο μαζί μας για να διασφαλιστεί η επάρκεια κονδυλίων για αυτό το πρόγραμμα. Αν υπάρξουν περικοπές από το Συμβούλιο θα πρέπει να επανεξεταστεί η θέση του Ευρωκοινοβουλίου και να συζητήσουμε τι θα κάνουμε αν υπάρξει σημαντική περικοπή από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Grazie la collega ε, ευχαριστώ. Συνάδελφο Έλερ έχει το λόγο. Τρία λεπτά. Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω κι εγώ και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την πολύ καλή δουλειά που κάναμε. Πολιτικά ε, καταφέραμε να έχουμε μια πλειοψηφία δύο τρίτων, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλή, δυνατή ε, ε, διαπραγματευτική θέση απέναντι στην Κομισιόν και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε. Κάποια σημεία τώρα, έτσι, τηλεγραφικά λόγω του σύντομου χρόνου που έχω. Σε πολλά μπορώ να συμφωνήσω με τις δύο κυρίες που πήραν το λόγο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου για την αριστεία, το Stairway to Excellence, είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα ότι η διεύρυνση του προγράμματος ό,τι αφορά τη συμμετοχή ε, από την Ευρώπη των 12 ε, την μπαίνει σε συζήτηση τώρα στο Συμβούλιο. Νομίζω ότι η πρόταση που έχει κάνει το Κοινοβουλίο, η πρόταση που έχει κάνει το Κοινοβούλιο είναι πολύ διαφοροποιημένη και σίγουρα θα πρέπει να την συνεχίσουμε να τη μελετούμε. Τώρα, για το ΕΛΚ υπάρχουν τρία-τέσσερα σημεία που θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι η αριστεία βεβαίω, το πιο σημαντικό κριτήριο. Το δεύτερο είναι μια ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού του ορίζοντα 2020 για τη διεύρυνση τη συμμετοχή. Το τρίτο είναι η ανεξαρτησία και η διεύρυνση μέσω επιπλέον ε, ε, μέτρων ε, για τα προγράμματα για τις ΜΜΕ. Και επίση το τέταρτο είναι η, σύνδεση με τα διαρθρωτικά ταμεία. Και θέλω να πω ότι αυτό έχει να κάνει και με το ότι υπάρχουν ε, ε, ε, κονδύλια από το ΕΦΡΙ που πρέπει να στοχοθετηθούν και να αποδοθούν εκεί που χρειάζεται. Είναι σημαντικό η κατανομή των απαιτήσεων αυτών να τις συμπεριλάβουμε σε δύο γραμμές του προπολογισμού. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ως προς αυτό. ούτως ή άλλως το Κοινοβούλιο θα λάβει ε, θέση και για τα δύο αυτά κομμάτια. Νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την έρευνα για την ενέργεια θα πρέπει να δούμε πάλι τον κατάλογο των μέτρων. Το ΕΛΚ εδώ έχει, κάνει κάποιες, ε, έχει υποβάλει κάποιες τροπολογίες ε, για την αποτελεσματικότητα, για το CCS, για τις μειώσεις των των εκπομπών των διοξιδίων του άνθρακα, το εναντοχή των ε, ευρωπαϊκών ε, εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας και επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ. Γι' αυτό έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις, οι οποίες γενικώ έχουν τύχει καλής υποδοχής. Βεβαίω πρέπει να τονίσουμε και το θέμα των διαγωνισμών, τη πρόσκληση υποβολής ε, προτάσεων, ενδιαφέροντο. Και για, τον συνολικό, για τη συνολική πρόταση του για τον ορίζοντα πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με μέσα και πρέπει να δούμε και το fast track to innovation ε, το οποίο θα πρέπει να, έχει να, αποτελέσει ένα συγκεκριμένο μέτρο έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τα ε, μέτρα προ, ε, έρευνας για τον ορίζοντα. Σημαντικό επίσης είναι η συμφωνία που έχουμε. Όλα πρέπει να πάνε πολύ πιο γρήγορα Σημαντικό επίσης είναι η ε, συμφωνία που είχαμε για την ε, τεχνολογία και για τα open course που θέλουμε να γίνουν και επίσης σημαντικό είναι ότι το, το πρόγραμμα στο σύνολό του είναι πολύ φιλικό προς τις καινοτομίες δεν ε, θέτει συγκεκριμένα άτεκτα ε, ε, στοιχεία, αλλά έχει μια, ένα βαθμό ευελιξία. Και ένα τελευταίο σημείο, η εφαρμογή των δημοσιονομικών μέσων. Πρέπει να συζητηθεί το θέμα αυτό εντατικά. Μιλούμε για 20 δισεκατομμύρια. Επί τη αρχή το χαιρετίζουμε, αλλά η πρικοδότηση αυτή νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει παραμείνει εκρεμέ και πρέπει να αποτελέσει κομμάτι τη συζήτηση που θα κάνουμε με την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος Γιωχάνσεν που δεν μπορεί να παραστεί γιατί έχει πάει με μια αντιπροσωπεία της ΣΤΟΑ στο Κιώτο. Εξ του κυρίου Γιώχανσεν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μαντουρέλ και την κυρία Καρβάλιο για την πολύ καλή δουλειά και την πολύ καλή συνεργασία. Ο κύριος Γιώχανσεν είναι αρκετά ικανοποιημένος με την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων μέχρι τούδε ένα ή δύο πράγματα όμως υπάρχουν που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Θα ανέφερα από αυτά τρία συγκεκριμένα ένα προς ένα. Πρώτον, η επικέντρωση στην ανάγκη της, ε, στις ανάγκες καινοτομίας και έρευνας που πρέπει να διασφαλιστεί. Κάπως ανησυχούμε, κάποιες πολιτικές ομάδες θέλουν να μεταθέσουν την επικέντρωση αυτή σε προανταγωνιστική έρευνα και να καταστεί αυτή η πτυχή ε, προτεραιότητα. Αν θέλουμε να διασφαλίσουμε με σοβαρό πνεύμα την αηφορία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το input στην έρευνα και ανάπτυξη θα δίνει πραγματικό output. Είναι σημαντικό θέμα η καινοτομία για την έρευνα και πρέπει και αυτό να αντανακλάται έτσι στο πρόγραμμα. Δεύτερον, η διεύρυνση συμμετοχής. Να διευρυνθεί η συμμετοχή γεωγραφικά είναι σημαντική υπόθεση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να το κάνουμε αυτό χωρίς να διακυβεύεται η αρχή της αριστείας γιατί διαφορετικά θα γίνει ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα απλώς αυτό. Ένα άλλο σημείο. Το 2020 δεν αφορά μόνο την αριστεία στην έρευνα αλλά και την αριστεία στην καινοτομία και στις δραστηριότητες σε σχέση με τις αγορές. Αν υπάρξει μετάθεση για παράδειγμα Πολλές φορές έχουμε και την συμμετοχή σε υπεργολαβίες Μία θηγατρική, για παράδειγμα, στη Σλοβακία θα μπορούσε να εξαρτάται από την έρευνα στη Γερμανία, άλλη από έρευνα στην Ισπανία. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα συζητάμε την διεύρυνση συμμετοχής. Και τέλος, ε, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην ομάδα μας, στην ομάδα, θεωρούμε ότι με ένα σφιχτό προϋπολογισμό ήδη σήμερα δεν θα πρέπει να κατακαιρματίζουμε τα θέματα και να διαχωρίζουμε τις προτεραιότητες και να έχουμε μια ξεχωριστή αντιμετώπιση πρόκλησης όσον αφορά την ασφάλεια. Αν υπάρξει ο κατακαιρματισμός αυτός θα χάσουμε την επικέντρωση από τις σωστές προτεραιότητες και θα έχουμε θέματα στρατιωτικά και άμυνας αποκλειστικά. Η συνέπεια ποια θα είναι θα είναι δυστυχώς ότι λιγότερα κονδύλια θα δαπανώνται σε σημαντικούς τομείς όπως την αποδοτικότητα για την ενέργεια, τα θέματα του, του κλίματος και των κλιματικών αλλαγών, τις περιβαλλοντικές πτυχές που είναι τόσο σημαντικές και σε σχέση με έναν ε, προϋπολογισμό που αντιμετωπίζει ήδη πιέσεις εξ ονόματος της ομάδας Άλντε θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να ληφθούν αυτά τα θέματα υπόψη. Ευχαριστώ. Grazie, la parola al signor Lambert. Ο κύριος Λάμπερς. Να επικεντρωθώ στα όσα είπε η Μαρία και η Τερέζα και στις εκθέσεις τους. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Ξεχνάω το όνομά σας στο μικρό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω το εξή. Δεν ε, δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να πάμε σε πολύ αυξημένο προπολογισμό. Ελπίζω να καταφέρουμε και μιλώ σε σένα τώρα, Κρίστιαν. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν θα έχουμε το, τον προπολογισμό που θέλουμε. Το να προσθέτουμε συνέχεια νέε δαπάνε είναι λίγο τρελό. Α, χαίρομαι που λε όχι. Εντάξει. Ε, Ειλικρινώ λοιπόν αυτό το θέμα είναι θέμα εθνικών προπολογισμών. Δεν μπορούμε απλώ να είμαστε εμεί μια διαδικασία διορθωτική στου εθνικού προπολογισμού. Βεβαίω εγώ θέλω να δω τι θα γίνει και με, τον, με την μεταφορά του, ευρωπαϊκού, του των κονδυλίων στον ευρωπαϊκό προβλεψμό από την άμυνα. Τότε θα είμαι ευχαριστημένο μόλι δω το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, για την έρευνα και την καινοτομία συμφωνώ με αυτό που είπε η Φιώνα. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Η Ευρώπη θεωρείται ότι είναι καλή προς τα πάνω, αλλά δεν καταφέρνει τελικά να έχει κέρδος. Δεν λέω βέβαια να πάμε μόνο στην, να αφήσουμε τελείως την έρευνα και να πάμε μόνο στην ε, πρακτική, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία δουλεύουν καλά σε ό,τι αφορά την κοινοτομία. Ε, Α πούμε το εργαλείο για τις ΜΜΕ, το Equity and Debt Facility, ε, θα μπορούσαν ίσως αυτά να αποτελέσουν την αιχμή του δώρατος. Και θα πρέπει όντω να έχουν και κατάλληλη πρικοδότηση. Ε, ξέρετε ότι εγώ θέλω να έχουμε έναν φιλόδοξο προπολογισμό για το εργαλείο για τις ΜΜΕ, γιατί ξέρουμε ότι δουλεύει καλά. Και επίση πιστεύω ότι αυτό είναι ο δρόμο όπου γίνεται όντω, αυτό είναι το μέσο που γίνεται όντω η καινοτομία. Επίση, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε προσθήκη στο JTI. Ε, ακόμα δεν έχω βρει, δεν έχω βρει έναν εμπλεκόμενο φορέα στο, στην, ε, ε, έρευνα και την καινοτομία πλην των, GT, που να μου πει χρειαζόμαστε αυτό το εργαλείο. Λυπούμε. Όλοι λένε αν πρέπει να ε, σκοτώσουμε μια ιερία γελάδα, αυτή πρέπει να είναι. <coughs> και για τα PPPs ε, είμαι πολύ περισσότερο υπέρ του να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε ένα ε, κομμάτι στο μοντέλο που, ε, χρηματοδότησης που θα, ε, ουσιαστικά θα υποχρεώνει τους επενδυτές να επενδύσουν παρά να συνεχίσουμε να προχωρούμε στον δρόμο που έχουμε ξεκινήσει γιατί δεν είναι σωστός. Πραγματικά λοιπόν πολλές, πολλά, πολλοί αστερίσκοι για τα PPPs. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν και άλλες, και άλλες οδοί για τα εργαλεία, εάν τελικά για να καταλήξουμε μόνο σε αυτό που προτείνεται. Δύο τρίτα της, ε, του προπολογισμού θα πάνε στην ε, έρευνα. Νομίζω ότι στην επόμενη περίοδο δεν θα πρέπει να μειώσουμε το ποσό αυτό. Οπότε εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Για τον ε, προπολογισμό, είπαμε ότι πρέπει να περιμένουμε ένα μεγάλο προπολογισμό, αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, προφανώ θα πρέπει να, κλείσουμε, να, μειώσουμε κάποιε από τι προκλήσει μα. Πρέπει δηλαδή να θέσουμε κάποιε προτεραιότητε. Αν η μείωση είναι 10-20%, προφανώς θα πρέπει κάποια projects να μείνουν λίγο πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ ίδια θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία που είχα μέχρι σήμερα για, αυτό το χαρτά, για αυτά τα χαρτοφυλάκια και για τη συνεργασία για τις τροπολογίες από τις διάφορες ομάδες είναι ένα καλό ε, σήμα για την κοινή μας συνεργασία. Θέλω απλά να αναφερθώ σε κάποια θέματα που θεωρώ ότι δεν έχουν κλείσει απόλυτα και πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα είναι απόλυτα αναγκαίο να καταλήξουμε σε συμφωνία σε σχέση με το ανοιχτό παράρτημα, την ανοιχτή πρόσβαση, open access, ανοιχτή πρόσβαση και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε, να συνεισφέρουμε με το πιο αποτελεσματικό τρόπο ως Ευρωκοινοβούλιο. Και είναι αναγκαίο να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, κάποιες προσαρμογές. Και συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε υπέρ του προϋπολογισμού για την επάρκεια των κονδυλίων. Και για την έρευνα και την καινοτομία δεν μπορούμε να συζητάμε για τέτοιου φιλόδοξους στόχους και μετά να έχουμε περικοπές από πλευρά του Συμβουλίου θα πρέπει να έχουμε μια στεναρή στάση για τη διασφάλιση των κονδυλίων αυτών. Τρίτον, πρέπει να πω ότι συμφωνώ ότι δεν πρέπει να έχουμε διευρύνσεις και άλλες εξαιρέσεις όσον αφορά τις δημόσιες και ιδιωτικές συμπράξεις, ΣΔΙΤ. Συμφωνώ σε σχέση με τον προλαλήσαντα συνάδελφο με την κυρία Λάμπερτα. Πρέπει επίσης να ε, υπάρξει ένα συμβιβασμό, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ε, κάποια τέτοια τάση. Για τα θέματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί σύμφωνο και έχουμε μια διεργασία που είναι πολύ επικοδομητική και ενδιαφέρουσα. τέλος, και ε, επειδή ε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, εδώ στην δυνατότητα εξέτασης αυτών των θεμάτων για τη χρηματοδότηση, χρηματοδότηση των πινάκων που έχουν παρουσιαστεί, που έχουν κατατεθεί όσον αφορά καταλόγων ή πινάκων, όσον αφορά τα θεσμικά όργανα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, επιχειρήσεις. Για τα δύο πρότυπα που προτάθηκαν από πλευράς του συναδέφου για τις ε, δράσεις ε, για την ανάπτυξη και την έρευνα, και για την ε, έρευνα σε σχέση με την ε, αγορά περισσότερο που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες ε, των επιχειρήσεων. Έχω αμφιβολίες για το πρότυπο που παρουσιάστηκε. Μπορώ ακόμα και να πω ότι θεωρώ χωρίς καμιά δυσκολία ότι η πρόταση που έκανα δεν γίνεται δεκτή, οπότε θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Αλλά πρέπει πρώτα να δούμε ότι υπό το κόστος που θα είναι επιλέξιμο θα πρέπει τα κέντρα ερευνών των πανεπιστημίων να έχουν πρικοδοτηθεί με τα ίδια μέσα όπως και οι βιομηχανίες και οι επιχειρήσεις. Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι μια σοβαρή προσέγγιση ή σωστή προσέγγιση, γιατί είναι τελείως διαφορετικές ε, οι μορφές και οι φύσεις των κονδυλίων στις, ε, στα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων και τα ερευνητικά κέντρα των επιχειρήσεων. για την πρόταση του 70% σε σχέση με την χρηματοδότηση, μπορώ να πω ότι ε, για το 70% μπορούμε να λάβουμε υπόψη μια τέτοια προοπτική. Αλλά υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν νέα κονδύλια, πώς θα υπάρξει δυνατότητα να προσληφθούν νέοι ερευνητές ε, με αυτό το πρότυπο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα έχουμε κόστη και μισθούς ε, σε σχέση με τους ε, ερευνητές που ήδη εργάζονται εκεί. Το περιθώριο λοιπόν που υπάρχει όσον αφορά την διεύρυνση του κόστους με την πρόσληψη νέων ερευνητών και μάλιστα νεότερων ερευνητών πάβει πλέον να υπάρχει. Αυτό θα ήθελα να εξετάσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε με το πρώτο μέρος. Πάμε για δύο λεπτά. Συνάδελφος Τζόρνταν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα απλά να απαντήσω σε αυτά τα οποία ακούσαμε ως παρατηρήσεις και σχόλια σήμερα. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω για άλλη μια φορά αυτό το οποίο επαναλαμβάνω κάθε φορά όταν συζητάμε για τον ορίζοντα 2020 ως θέμα. Θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει μια πιο ίση κατανομή κονδυλίων από την κατανομή που διασφαλιζόταν από πλευρά κονδυλίων στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Η πρώτη και κυριότερη προτεραιότητα πρέπει να είναι η επιστημονική αριστεία. Όμω, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε συνέργειες πρέπει να έχουμε κάποιε ευαισθησίε για κάποια θέματα. Ιδιαίτερα για το ότι οι ερευνητέ θα πρέπει να έχουν ίσες ισότιμες ε, προϋποθέσεις εργασίας για την έρευνά τους και την εργασία τους. Έχω δύο προτάσεις που θα τις δείτε σε τροπολογίες. Ε, πρώτον, αυτά θα πρέπει να αντανακλώνται και στους μισθούς, ε, στις απολαβές που θα έχουν υπό αυτό το πρόγραμμα οι ερευνητές. Θα πρέπει το ίδιο αντίτιμο, το, οι ίδιες ε, ε, ας το πω παροχές να λαμβάνονται υπόψη και να παρέχονται λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος διαβίωσης. Ε, και οι ευρωβουλευτές έχουν ισομισθό και φορολογούνται διαφορετικά ανάλογα με τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει και να λάβουμε υπόψη και το κριτήριο του, της αποδοτικότητας κόστους-οφέλους. Και πάλι εδώ, σε σχέση με τους αξιολογητές και την αξιολόγηση, πολλές φορές ακούμε ότι είναι δύσκολο να έχει κανείς πρόσβαση σε κάποιο τέτοιο δίκτυο. Πρέπει να υπάρχει μια νομοθετική πρόταση λοιπόν που θα διασφαλίζει τον ανοιχτό χαρακτήρα Υποστηρίζω τα πάντα, όλα όσα αναφέρθηκαν για την απλούστευση, για ένα βελτιωμένο, μια βελτιωμένη αναλογία ε, μεταξύ μεγαλύτερων και μικρότερων τέτοιων σχεδίων και προγραμμάτων για την έρευνα, καθώς επίσης και την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπό το σημερινό πλαίσιο η αναλογία αυτή θα πρέπει να είναι, είναι 15% και θα πρέπει να παραμείνει η αναλογία αυτή και να συνεχίσει να ισχύει και να υπάρχει δυνατότητα και σε μικρές επιχειρήσεις να συνδέονται και θα πρέπει να συνδέονται οι μισθοί και οι απολαβές περισσότερο με τις ε, απο, ε, που ε, παρέχονται και καταβάλλονται στις επιχειρήσεις σε σχέση με πανεπιστήμια θα πρέπει να προτείνουμε ένα τέτοιο πρότυπο γιατί είναι το μόνο το οποίο διασφαλίζει τη διασύνδεση μεταξύ εκπαίδευσης, παιδείας, καινοτομίας, κατάρτισης και έρευνας. Ευχαριστώ κύριο Ζιδάκου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο οι προλελήσαντες δεν ανέφεραν. Συμφωνώ με την κυρία Ριέρα ότι χρειάζεται ευεφία για στην αντιμετώπιση του, θέμα του θέματος της πρόσβασης στην πληροφόρηση. Διότι όταν έχουμε πρόσβαση στην πληροφόρηση έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Διότι όταν η πληροφορία τρέχει τότε και νέες ιδέες δημιουργούνται και νέα προϊόντα εμφανίζονται. Απ' την άλλη μεριά επίσης οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μείνουν χωρίς τα δικαιώματά τους. Οπότε ούτε όλα πρέπει να είναι δημόσια, ούτε τα αποτελέσματα της έρευνας θα πρέπει να είναι κλειστά μέσα σε ένα γκέτο και να μην βγαίνουν ποτέ. Πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία. Εγώ τόνισα ορισμένα ζητήματα που θεωρώ ότι είναι ενδιαφέροντα να έχουμε μία πολυεπίπεδη εστίαση διότι έχουμε διατομεακές έρευνες που μας δίνουν αποτελέσματα Και θα πρέπει επίσης να γίνουν σεβαστές οι αρμοδιότητες των εντεταλμένων πράξεων για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε κάποιες επιφυλάξεις, διότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα στον κόσμο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτόν τον τομέα. Ο κύριο Τσουκαλάς. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Τσουκαλά. Το μικρόφωνο του κυρίου Τσουκαλά παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συναδέλφους που μίλησαν πριν. Βρίσκω ότι σε αυτό το επίπεδο της συζήτησης, το γενικό επίπεδο της συζήτησης, αισθάνομαι την υποχρέωση να τονίσω δύο-τρία πράγματα. Το ένα είναι το ύψος της σημαντικής χρηματοδότησης. Είναι αδύνατο να φανταστώ αυτά που κυκλοφορούν ως φήμες. Ότι δηλαδή ο ορίζοντας 2020 επεξεργασμένος με φιλοδοξία θα προσγειωθεί σε αριθμούς οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη φιλοδοξία να φαίνεται μόρο φιλοδοξία. Εάν αυτό συμβεί, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξανααποδείξει ότι δεν πιστεύει σε αυτό τον τύπο της ανάπτυξης, δηλαδή στην ανάπτυξη που στηρίζεται στην έρευνα και την τεχνολογία. Σας παρακαλώ να σημειώσετε ότι ο ίδιος καυγάς γίνεται αυτό τον καιρό στην Αμερική, ακριβώς στην προεκλογική περίοδο με την αναγγελία ότι θα, κουπούν, θα περικοπούν 12 δισεκατομμύρια από τη χρηματοδότηση του NSF κοντεύει αυτό το ζήτημα να ανατρέψει τις αμερικάνικες εκλογές. Το δεύτερο σημείο είναι το open access, η ανοιχτή πρόσβαση. Θεωρώ ότι γίνεται μία συζήτηση κυριολεκτικά στο βρόντο. Αυτό το ζήτημα είναι λιμένο, δεν είναι τόσο περίπλοκο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το μπλέκουμε τόσο πάρα πολύ. Νομίζω ότι η κυρία Καρβάλιο και η κυρία Μαντουρέλ έχουν φτάσει σε μία συμφωνία η οποία κατοχυρώνει την ασφάλεια των αποτελεσμάτων των ερευνητών, την ταχύτητα και την δημοσιότητα των αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα και στο κοινό και καθιερώνει την απαραίτητη προϋπόθεση ο πολίτης να ξέρει πού πήγαν τα λεφτά του. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά τα ευχαριστήρια και τα συγχαρητήρια στους εισηγητές και θέλω να επιμείνω σε ένα σημείο που νομίζω η κυρία Καρβάλιο το έθιξε η συγκυρία που είναι βασικότατη αφορά στην ψηφοφορία για το πολιετές πλαίσιο. Στις 23 του μηνός έχουν ένα συμβούλιο που περιμένουμε να δούμε τι θα βγει για τον ΕΚΕ. Την επόμενη ψηφίζουμε στην Ήτρε μετά την Ολομέλεια του Στρασβούργου ο Πόη θα θέσει μία πρώτη πρόταση εκ μέρους του Συμβουλίου και θα ξέρουμε προς τα πού πάμε. Αν η πρόταση είναι μία περικοπή όχι πολύ μεγάλη, ας πούμε ένα 10% τότε μπορούμε να έχουμε μία κατανομή. Αλλά αν η πρόταση είναι πολύ μεγαλύτερη τότε πρέπει οπωσδήποτε να αποφασίσουμε για τις προτεραιότητες. Είναι θεμελιώδες. Και αυτό που ζητώ από τους εισηγητές, λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή ότι μετά το Στρασβούργο έχουμε την πράσινη εβδομάδα και μετά φτάνουμε πια στο Νοέμβριο, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μία μονογραφική συζήτηση για αυτό το θέμα. Όταν δηλαδή τελειώσει η Ολομέλεια και θα ξέρουμε και ποια είναι η πρώτη πρόταση που θα διατυπώσει το Συμβούλιο μέσω του Προέδρου του. Κύριος Βανίστερόη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να κάνω μια παρατήρηση, θα ήθελα πρώτον. Όταν υπάρχει κάποια επίθεση θα πρέπει έγκαιρα να διασφαλίζει κανείς την άμυνα και το τι θα κάνει. Δεύτερον, για τα κόστη τα οποία θα πρέπει να καλυφθούν και για την έρευνα και για το 2013. Και θα πρέπει εδώ να δούμε ποια προγράμματα θα υπάρξουν όχι να μην υπάρχουν κονδύλια μετά στη συνέχεια ώστε τέτοια ε, προγράμματα να χρηματοδοτούνται. Θα πρέπει οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί να εξοφλούνται και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012. Στον προϋπολογισμό του 2013 αν υπάρξουν περαιτέρω ε, περικοπές θα υπάρξει φθήνουσα πορεία και δεν θα πάμε καθόλου καλά αυτή είναι η κλίμακα που θέλουμε να ακολουθήσουμε για την αριστεία. Και βλέπουμε τώρα εδώ τους εισηγητές που ασκούν πιέσεις για να βελτιωθούν τα πράγματα και το εκτιμώ αυτό. Πρέπει να δούμε πώς τα κονδύλια για τον ορίζοντα 2020 θα μπορέσουν να τύχουν τις σωστότερες χρήσεις και να διασφαλιστούν κιόλας με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε και τις χώρες συνοχής, έχουμε τα διαφορετικά ταμεία, το Ταμείο Συνοχής και Σύγκλησης και θα πρέπει εδώ τα κονδύλια αυτά να μπορούν να έχουν ε, την καλύτερη χρήση για τον της δημοκρατική, την δημοκρατική αλλαγή, τον εκδημοκρατισμό, για το νέο συμβιβασμό 3 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν προγράμματα για την ενεργό για την ε, ε, υγεία των πολιτών, ε, να μην αμεληθούν αυτά. Ζητώ υποστήριξη λοιπόν ώστε αυτοί οι τομείς να καλυφθούν επαρκώς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ άκουσα όλα όσα είπαν οι συνάδελφοί μας μέχρι σήμερα και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Και εκφράζω τη βαθιά ανησυχία την οποία τρέφω. Διότι εδώ και χρόνια εμείς εκτιμούσαμε ότι αυτό το οποίο χορηγείται στην έρευνα ήταν ανεπαρκές και σήμερα φτάσαμε να αναρωτιόμαστε τι θα απομείνει μετά τις διαπραγματεύσεις. Υπάρχει ένας τομέας πολύ σημαντικός για την έρευνα, είναι ο τομέας της υγείας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στους πολίτες μας. Η μεταρρύθμιση στον τομέα της υγείας είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούν ιδιαίτερα οι πολίτες. Εγώ δεν θα πάρω ε, σημείο προς σημείο το τι προτείνεται εδώ για την υγεία. Θέλω απλώς να σας θυμίσω πόσο είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συντονισμός του συστήματος παρακολούθησης, του συστήματος συναγερμού, της παρακολούθησης των αλλαγών στον τομέα της υγείας. Χρειάζεται δηλαδή να καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες στον τομέα της έρευνας. Χρειαζόμαστε διατομεακές προσεγγίσεις δηλαδή μέσα εμπίπτουν τα μαθηματικά, η φυσική, η πληροφορική, είναι κάτι το πολυεπίπεδο η έρευνα στο ιατρικό τομέα. Υπάρχει το θέμα της επένδυσης, ε, των επενδύσεων στις νανοτεχνολογίες και στις ευρυσιτεχνίες. Θα ήταν κρίμα να εγκαταλείψουμε αυτόν τον τομέα στους Ασιάτες ή στους Αμερικάνους. Και δυστυχώς η Ευρώπη να χάσει ένα στάδιο που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Γκουτιέρες Κορτίνες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές για τον τρόπο που εργάστηκαν, άκουσαν τους πάντες και θέλαν να καταλήξουν σε μία ενιαία θέση. Επεξεργάστηκαν ένα κοινό σχέδιο πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους και την Τερέζα Ριέρα και τους άλλους. Θέλω όμως κάτι. Ε, χαίρομαι για την ενίσχυση των, του πολιτισμού. Απ' την άλλη μεριά όμως επιμένω ότι πρέπει να αλλάξουμε τα θεσμικά μοντέλα δίκησης και διαχείριση των πόρων. Ρωτώ, τι γίνεται με τα μικρά σχέδια. Διότι η Ευρώπη μιλάει εδώ για μεγάλα σχέδια, 5 εκατομμύρια ευρώ, 9 εκατομμύρια ευρώ, αλλά με τα μικρά σχέδια τι γίνεται, που είναι αυτά δηλαδή που, με τα οποία ασχολούνται τα περισσότερα πανεπιστήμια και δεν απαιτούν τόσο μεγάλα κονδύλια. Και για την multi-research, είναι σχέδια τα οποία δεν έχουν καν ερευνητέ μέσα μερικά από αυτά και είναι χαμηλής ποιότητας. Και τώρα που διαλύεται όλο το σύστημα και εξωτερικοποιούμε την Γενική Διεύθυνση Έρευνας, πώς θα λειτουργήσει η αριστεία και η συνέργεια που βρίσκεται. Διότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα σωρό τροπολογίες για τα διαρθρωτικά ταμεία. Πώς προχωράμε, τι γίνεται. Κύριος Πρόντι. Εγώ, Πρόεδρε, ήθελα να σταθώ σε ένα τμήμα του προϋπολογισμού που βάζει μαζί την Ήτρε με τον Γαλιλαίο και το GMS. για διακυβερνητική διαχρηματοδότηση. Το ίδιο όμως είναι ένα πρόγραμμα καθαρά ερευνητικό και δυστυχώς δεν έχει ακόμα εφικτά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να συνεχιστεί. Ενώ τα προγράμματα Γαλιλαίος και GMS μοιάζουν με διαρθρώσεις που είναι πραγματικά ευρωπαϊκές και πρέπει να συμπληρωθούν το νωρίτερο δυνατό για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να, μην, να αφαιθεί έτσι στη διακυβερνητική πρωτοβουλία, αλλά να υποστηριχθεί από τα κοινοτικά ταμεία. Κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις έγιναν και συμφωνώ με αυτές. Το κυριότερο σημείο είναι ότι έχουμε τον ορίζοντα 2020 και πρέπει να δούμε την, ε, το ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και δεν πρέπει να αμελήσουμε αυτή την αναλογία. ορίζοντα ορίζοντας 2020 που αρχικά είχε 100 δισεκατομμύρια, τώρα έχει 80 δις, πρέπει να επανέλθουμε στα 100 δις με την βάση της, ε, των δραστηριοτήτων που θέλουμε να καλύψουμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει μια φθήνουσα εξέλιξη. Δεύτερο θέμα ιδιαίτερη σημασία και αυτό είναι ότι η έρευνα και η καινοτομία δεν μπορούν να αγνοηθούν σε σχέση με συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να δούμε για παράδειγμα και σε σχέση και με την ε, ε, ε, τα ανανεώσιμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα που θα πρέπει να οδηγεί σε καινοτομία. Αυτό πρέπει να είναι η κλειδί η κλειδί που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη, σε παραγωγικότητα, στην επίτευξη περιφερειακών στόχων της στοχοθέτησης του ορίζοντα 2020. Σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρξει μια κατάσταση όπου θα υπάρχουν ερευνητικά ιδρύματα στην Ευρώπη που δεν θα ε, εντάσσονται μέσα σε αυτή την προσπάθεια σε σχέση με κονδύλια τα οποία θα έπρεπε να, να διασφαλίζονται για να προχωρεί η έρευνα. Πρέπει εδώ να πούμε ότι θέλουμε την έρευνα την καινοτομία που οδηγεί σε θέσεις απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της ύφεση. Πρέπει σε αυτές τις ιδέες να επικεντρωθούμε. Ευχαριστώ. Κολέγια Χέλμα, Χέλμα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, Παρακολούθησα τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Παρακολούθησα τη συζήτηση με ενδιαφέρον. Οι ψηφοφόροι μου στι East Midlands στο Ηνωμένο Βασίλειο με χαρά θα ακούσουν ότι το πρόγραμμα 2020 θα έχει και μια fast track ε, για την ε, ε, καινοτομία και την αριστεία. Διαρωτώ με σε σχέση με την περίοδο αυτή των προϋπολογισμών για τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλα θέματα που πιέζονται ιδιαίτερα υπό τη σημερινή συγκυρία, αν θα κατανοούσαν οι ψηφοφόροι μου την ανάγκη του ότι θα πρέπει να τονίζεται η μεγιστοποίηση των κονδυλίων για αυτό το πρόγραμμα. Κάνουμε λόγο για ένα πολύ μεγάλο ποσό χρηματικά, αλλά αυτό το ποσό θα κατακαιρματιστεί και θα δίνεται σε αιτήσιες δόσεις και σε διάφορα κεφάλαια μεταξύ 27, 28 και κρατών μελών και πολλών θεσμικών οργάνων σε αυτά τα κράτη-μέλη. Και όσοι ήθιστε με οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πολλά από τη χρηματοδότηση θα απορροφηθούν για την αξιολόγηση, μελέτη κτλ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να προβληματιστούν να δουν αν αυτό το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο βέλτιστος τρόπος να επιτευχθεί η βέλτιστη ε, ωφέλεια σε σχέση με τα κονδύλια που δαπανούμε. Ή μήπως θα έπρεπε να υπάρξει κατανομή κονδυλίων ή επικέντρωση στα κράτη-μέλη περισσότερο. Και να πούμε ότι δεν πρόκειται τόσο πολύ για την καινοτομία και την έρευνα, αλλά για την ε, ας το πω έτσι, ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιου τομείς, από τους οποίους έχουν κάποιοι συγκεκριμένα ωφέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, πρέπει να πω επίσης σε όλους τους εισηγητές ε, και τους συναδέλφους ε, που υποστήριξαν τις τροπολογίες μου θα ήθελα να επικεντρωθώ στα εξής τρία σημεία που ακολουθούν. Πρώτον, ο λόγος, η αιτιολογία για την διασύνδεση της επιχειρηματικής και ερευνητικής σφαίρας μπορεί να λειτουργήσει όταν υπάρχουν κονδύλια. Μόνο όταν υπάρχουν επαρκή κονδύλια μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια συνάρτηση. Τώρα με τον ορίζοντα 2020 παρέχεται μια θετική, καλή βάση για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεύτερη παρατήρηση. Στις τροπολογίες συμπεριλάβαμε την καινοτομία σε τομείς όπως ορεινές περιοχές και θαλάσσιες περιοχές παράκτιες περιοχές. Πολλές φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και ε, εγκυμονούν εδώ σε αυτούς τους τομείς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Τρίτον, σε σχέση με την ιατρική, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ηλικιωμένους, τους υπερήλικες ε, που έχουν υποστεί και κάποια εγχείρηση, φροντίδα και περίθαλψη που θα πρέπει να δίνεται. Θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες για τηλεπαρακολούθηση και τηλεπαροχή τέτοιας περίθαλψης. Η κυρία Τικάου παρακολουθεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ από πλευράς μου τους εισηγητές και τις εισηγήτριες. Ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκαν είναι εξαιρετικός. Πρέπει να πλουστεύσουμε τις διεργασίες. Ο ορίζοντας 2020 είναι μια απλουστευμένη στρατηγική για τα θέματα έρευνας, για τα προγράμματα έρευνας και αυτό είναι καλοδεχούμενο. Επίσης, χαιρετίζω την επιλεξιμότητα προγραμμάτων στον τομέα όσον αφορά τις δημογραφικές αλλαγές, περιβαλλοντικές αλλαγές, περίθαλψη στον τομέα της υγείας, ε, υγειονομική περίθαλψη κτλ. Ως προς αυτά θα ήθελα να πιστήσω την προσοχή σας σε κάποιες τροπολογίες που έχω καταθέσει. Προσπάθησα από πλευράς μου να δώσω ένα πιο ευδιάκριτο ρόλο και χαρακτήρα ε, ε, στα προγράμματα επίδειξης και πιλωτικά προγράμματα στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή στον τομέα της γεωργίας δίνοντας δυνατότητα σε σχέση με κονδύλια που θα παρέχονται που θα καλύπτουν 100% τα κόστη επιλεξιμότητας. Θα έλεγα ότι λαμβανομένων υπόψη όλων αυτών τα κονδύλια που πληρώνονται για παράδειγμα για έναν μισθό ε, αναώρα, ένα ποσό που καταβάλλεται αναώρα, θα πρέπει να είναι όμοιο ένα τέτοιο ποσό για τα διαφορετικά κράτη-μέλη και θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή των επιχειρήσεων και έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η έρευνα δεν θα μένει σε ένα ε, κλειστό στεγανό πλαίσιο, θα έχει πρόσβαση στην αγορά και θα έχει πρόσβαση στους καταναλωτές και αυτό θα είναι μια δυνατότητα να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Η τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να αναφέρω είναι η διαδικασία επαναβιομηχανοποίηση στην ε- Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μια άμεση, ένας άμεσος συσχετισμός, μια άμεση αναλογία μεταξύ έρευνας ε, και ανάπτυξης για την ε, επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας τη δυνατότητα σε αυτή τη δυνατότητα των βιομηχανιών να είναι ανταγωνιστικές στην σε παγκόσμια κλίμακα. Μόνο έτσι μπορεί να είναι ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης και τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις και να είναι θετικό αυτό για το τι θεωρούμε σημαντικό από πλευράς μας. Ακούω επανειλημμένα και αναφέρεται διαρκώς ότι πρέπει να τεθούν κάποια κεντρικά σημεία, κάποια κέντρα βάρους. Εντάξει, όμως πρέπει να δούμε ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ημερομηνία ψήφισης προς έγκριση και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Έχουμε τώρα θέματα προσωπικών επιλογών και προτιμήσεων. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και πιέζει ο χρόνος. ριούμενε τι και θα πρέπει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Ακούμε επίσης ότι το Συμβούλιο έχει υπόψη του να περικόψει και μάλιστα κατά το ίμιση τα κονδύλια αυτού του ε, τομέα. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί και να μας δημιουργήσει προβλήματα, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τέτοια προσέγγιση. Συνάδελφοι, πρέπει παρακαλώ συγκεκριμένα να δούμε τι θα κάνουμε, με συγκεκριμένα προγράμματα για τον προϋπολογισμό, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και μια τελευταία παρατήρηση. Έχω την εντύπωση που αποκόμισα ότι πάντα και επανειλημμένα επικεντρωνόμαστε στην έρευνα. Αλλά εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας. Θα πρέπει εδώ να δούμε και την μετάθεση στην καινοτομία. Δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Πρέπει πολύ συγκεκριμένα και εξειδικευμένα να προβληματιστούμε, να τα συλλέξουμε, να τα συμπτύξουμε, να τα συνενώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να είμαστε αποτελεσματικοί. Να μην είμαστε, να μην κατακαιρματιστούμε, αλλά να συμπυκνωθούμε και να συμπτύξουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Οντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια για τα μεγάλα σχέδια, Ήτερ, Γαλιλαίο, GMS. Αν κατάλαβα καλά όσα είπε ο κύριος Πρόντι, είναι να διαχωρίσουμε το τι είναι κοινοτικό, ας πούμε ο Γαλιλαίος και τα άλλα να τα ε, διακυβερνικοποιήσουμε. Δεν πρέπει όμως να βγούμε από την ευρωπαϊκή λογική. Θα ήταν μια ευρωπαϊκή άρνηση, απάρνηση και δεν θα έλυνε τίποτα το ίτερ. Δεν είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο, είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο. Ποια θα ήταν η εικόνα που θα δίναμε αν δεν μπορούσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να προωθήσουμε το ίτερ για τα θέματα που συζητάμε. Εγώ ήμουν εισηγητής ε, για τα τέσσερα πρώτα χρόνια 25 δις ε, στα 51. Μας μένουν 30 εκατομμύρια για το 2000-2013 ε, για την έρευνα. για τον ορίζοντα 2020 εμείς χάνουμε την ευρωπαϊκή της έρευνας Και θα ήθελα στη ρήτρα αναθεώρησης το να φανταστούμε ότι θα διαπραγματευτούμε 100 δις έτσι όπως έχει κατάσταση σήμερα στα κράτη, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να αρχίσουμε να καυγαδίζουμε διότι άμα μαζέψουμε και τον καυγά για τη Γεωργία και το τα θέματα των Βρετανών, έχουμε και τις εκλογές στη Γερμανία, ρεζίλ θα γίνουμε ανά τον κόσμο. Πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να ανασάνουν, να ψηφίσουν, ναι, ό,τι είναι να ψηφίσουμε και μετά το 2016 όπου θα έχουμε συνέλθει και θα έχουμε και ένα νέο κοινοβούλιο να ζητήσουμε μία αναθεώρηση. Τώρα έχουμε λαμπρούς επιστήμονες αλλά για τη βιομηχανική ε, καθεδρία δεν λέμε τίποτα, η Κομισιόν δεν λέει τίποτα. Θα έπρεπε και αυτό να γίνει μία κοινωνική πρόκληση. Ο κύριος Μινίν. Στι Στις διάφορες ακροάσεις που κάναμε καταλάβαμε ότι ο καθένας είχε ένα μήνυμα. Αλλά εκείνο το οποίο καταλάβαμε επίσης είναι ότι η έρευνα είναι κάτι το πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα το ότι το καταλάβαμε είναι καλό. Άμα, είχαμε, άμα μας δίναμε και τις δυνατότητα να προχωρήσουμε μακρύτερα αυτό θα ήταν καλύτερο. Αν εμείς αντιπαραθέσουμε το μίσο όπως είναι η έρευνα ή όπως και την αντιπαραθέσουμε με την υγεία, τότε αποσταθεροποιούμε ένα ολόκληρο σύστημα. Εδώ τι έχει γίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε απαλλάξει φορολογικά κάτω το, το, το κεφάλαιο και δεν έχουμε προχωρήσει σε πράγματα χρήσιμα για την κοινωνία. Εμείς θα, θα, θα μπορούσαμε να κοιτάμε μόνο τον οφαλό μας. Αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι έτσι θα βρούμε τη λύση. Αν μάθουμε εμείς να, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, τι μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε ότι εμείς έχουμε μείνει πίσω, ότι οι Κινέζοι έχουν προχωρήσει, οι Ιαπωνέζοι έχουν προχωρήσει, οι Αμερικάνοι έχουν προχωρήσει. Θέλουμε να προχωρήσουμε, συνεχίσουμε να προχωράμε έτσι. Μίλησε ο κύριος Βανίστερο για ποδόσφαιρο, αλλά η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο ισχύει για την έρευνα. Πρέπει να επενδύουμε παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω για να ξεπεράσουμε τους αντιπάλους μας. Αυτό το οποίο κάνουμε, τι λένε, τι λέμε, Λέμε ναι, ναι, αυτοί όλοι οι άλλοι είναι πιο, πιο δυνατοί από εμά. Εμείς είμαστε οι πιο ανίσχυροι, οπότε ωραιότατα. Μειώνουμε τον προϋπολογισμό. Και να πάμε ακόμη χειλότερα. Πληρώνουμε όμως δισεκατομμύρια τους ποδοσφαιριστές για να τους παίρνουμε για μια ομάδα να βρίσκονται σε ένα γήπεδο και δεν πληρώνουμε τους ερευνητές που αποτελούν μια σημαντική πρόκληση για την Ευρώπη. Το να μην επενδύει κανείς σε κάτι το οποίο έχει μία άμεση αποδοτικότητα ε, είναι λάθος. Διότι οι επενδύσεις στην έρευνα είναι, και στην πολλαπλή έρευνα είναι αυτά που θα δώσουν αποτελέσματα και μετά πρέπει να παίζουμε συλλογικά. Διότι άμα παίζει ο καθένας μονάχος του στο δικό του γήπεδο δεν θα έχουμε ποτέ δύναμη. Κύριο Έλερ. Δύο άμεσες απαντήσεις να δώσω στην αντίρρηση των πράσινων και της Άλντε για το θέμα της έρευνας για την ασφάλεια και από πλευράς Λάμπερς για την ασφάλεια. Δεν είναι το θέμα του ΕΛΚ για την άμυνα. Αυτό το οποίο κάναμε και κάναμε από κοινού με την Άλντε, τους πράσινους τους σοσιαλιστές, το ΕΛΚ και άλλες ομάδες είναι προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε αυτά τα οποία αποφασίσαμε σε μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη για το πρόγραμμα έρευνα. Έρευνα για πολιτικούς σκοπούς και για στρατιωτικούς σκοπούς διτά, γιατί αποτελούν σημαντικές μορφές ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεύτερον, θέλω να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπε ο Ρότζερ, αν θα το κάνουμε αυτό σε εθνικό επίπεδο ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για φανταστείτε αγαπητέ Ρότζερ, η Rolls Royce, το μαργαριτάρι της ε, βιομηχανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν είχε ε, σε σχέση με το 70% ε, για την έρευνα. Στη δική μας ε, χώρα δεν είναι μόνο θέμα εθνικής βιομηχανίας. Έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη, ας οικονομία και επιχείρηση. Και πρέπει εδώ να δούμε τα θέματα αυτά. Έχουμε την Ευρώπη στην έρευνα δεν έχουμε το αντίστοιχο ενό προγράμματο, αλλά υπό πρακτικού όρου είναι η Ευρώπη που αναλαμβάνει την έρευνα και όχι πλέον τα κράτη-μέλη ή τα εθνικά πανεπιστήμια που επομίζονται αυτή την έρευνα για εθνικούς σκοπούς. Λοιπόν, υπό το δικό μου πρίσμα, ποια θα μπορούσε να είναι η επικέντρωση. Απεγνωσμένα αναζητούμε δυνατότητε ανάπτυξη και σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουμε μια σημαντική ε, πτυχή για την έρευνα, για την ανάπτυξη. Αν δεν επενδύσουμε θα μείνουμε πίσω. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να σημειώσουμε ανάπτυξη. Να μην ε, ομφαλοσκοπούμε στις συζητήσεις μας και να μην λαμβάνουμε υπόψη αυτά τα οποία γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα, αν θέλουμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη το δικό μας πρότυπο και το κοινωνικό μας πρότυπο πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα. Διαφορετικά θα ακολουθήσουμε μια φθήνουσα πορεία, δεν θα είμαστε σε θέση να είμαστε ανταγωνιστικοί. Αυτό πρέπει να κάνουμε και να δώσουμε από κοινού μάχη για τα κονδύλια του προπολογισμού, για τα δημοσιονομικά κονδύλια. Γιατί διαφορετικά δεν θα βρισκόμαστε σε ισότιμο επίπεδο, ας το πω έτσι, με τις ε, παγκόσμιες άλλες ε, δυνάμεις που εμπλέκονται σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ο Διευθυντής Ματέη εκ μέρους της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καθησυχαστικό να ακούω τους συναδέλφους εδώ, γιατί βλέπω ότι υπάρχει σύγκληση, η οποία σταδιακά επετεύχθη και πραγματικά τη χρειαζόμαστε. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει μία ενιαία θέση. Είναι πολύ δύσκολη η συζήτηση που θα γίνει συνολικά για τον προπολογισμό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, προβλήματα με τις πληρωμές, ε, με τις πιστώσεις πληρωμών. Το... Ξέρουμε πώς έχει λοιπόν η κατάσταση και έχουμε και τον ορίζοντα 2020 που αφορά πλήρω την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασία. Έχουμε κάνει την αξιολόγηση επιπτώσεων, είδαμε ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε 0,9 του ΑΕΠ επιπλέον λόγω του ορίζοντα 2020. Δεν είναι και λίγο. Ψέχνουμε να βρούμε για, την ισότητα των δύο φύλων ε, σύγκληση. Η κυρία Μαδουρέλη είπε ότι έχουν υπάρξει σαφεί γραμμέ. Έχουμε το open access, τη ελεύθερη πρόσβαση. Βεβαίω πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα δεδομένα, να το προσέξουμε πολύ. Και επίσης θα ξεκινήσει ένα πιλωτικό προγράμματα για, την, για θέματα IPR και εμπορικών συμφερόντων που θα πρέπει να διατηρηθούν. Επίσης, για τα βλαστοκύτταρα. Είμαστε ευγνώμονες που υποστηρίξατε το, την προσέγγιση αυτή για το status quo. Τώρα, είπατε κάτι για τη διεύρυνση της συμμετοχής. Η Κομισιόν ξέρετε ότι θέλει να δημιουργήσει έτσι, γέφυρες για, το, για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Έχουν υπάρξει πιλωτικά προγράμματα ε, πάνω στον τομέα αυτό και επίσης πρέπει να υπάρξει ένα μεγάλο φάσμα εργαλείων από τις διάφορες χώρες ώστε να μπορέσουν όλοι να βρεθούν στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, Ακούσαμε για το earmarking, την κατανομή κονδυλίων συγκεκριμένα, που ήταν πολύ σημαντικό. Βεβαίω υπάρχουν προτεραιότητε ω προ αυτό. Για την ενέργεια ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι τα διάφορα προγράμματα ανά χρονιά. Βεβαίω είναι μεγάλη πρόκληση αυτό. Η υγεία επίση είναι μεγάλος, ε, μεγάλη πρόκληση για κάθε α, πολίτη. Για την απλούστευση τώρα και τα ωφέλη των συμμετεχόντων. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικό που έχετε δώσει τόση σημασία έτσι ώστε ο ορίζοντα 2020 να επικεντρώνεται στον ε, όποιον συμμετέχει. Προφανώ πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ποιότητα όλη αυτή τη διαδικασία ε, σε, όλα τα, σε όλες τις φάσεις της. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και μια ευελιξία για τα εργαλεία αυτά, γιατί πρέπει να καλύψουμε μια ποικιλία ε, εμπλεκόμενων φορέων, ένα ευρύ φάσμα εμπλεκόμενων φορέων. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν οι ΜΜΕ, τι αναφέρατε όλοι, είπατε ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις ΜΜΕ και ναι, προτείνουμε νέα μέτρα ως προς αυτό, όπως ο, ο συγκεκριμένο μηχανισμός ε, για τις ΜΜΕ. Επίσης, ε, Έχουμε και προγράμματα για τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και γι' αυτό χρειαζόμαστε και ευελιξία για τα προγράμματα αυτά. Επίσης, ε, τα ΣΔΙΤ είναι σημαντικό θέμα, αν και λίγο αμφιλεγόμενο. Εκεί όντως πρέπει να προσέξουμε πολύ συγκεκριμένα τι έχει επιδευθεί και πρέπει να γίνει μια πολύ στέρεα αξιολόγηση επιπτώσεων έτσι ώστε να δούμε ποια θα ανανεωθούν, ποιες ε, συμπράξεις δημοσίου και δικού του θα, θα ανανεωθούν. Ε, ο κύριος ε, Έλερ επίσης ε, έχει δουλέψει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Έχουμε δει τα στοιχεία που προτείνονται. Οι επιδοτήσεις, ο χρόνος για, την απόδοσή τους θα είναι το μέγιστο δυνατόν. Η Κομισιόν έχει προτείνει μία πλούστευση και θεωρούμε ότι θα υπάρξει βελτίωση. Έχει υπάρξει και γνωμοδότηση επί του θέματος και το δικαστήριο λέει ότι το μοντέλο αυτό θα ε, βελτιώσει την αξιοπιστία του θα μειώσει το κίνδυνο παρατυπιών για τους, για τους επιλέξιμους φορείς, θα μπορέσει η όλη η λογιστική του πράγματος να γίνει πιο απλή και θα βελτιωθούν κάποια προγράμματα επαληθεύσεων που προκύπτουν από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, έτσι ώστε να βελτιωθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία εφαρμογής. Αυτά λέει το δικαστήριο. Είναι σημαντικό ότι ο ορίζοντας 2020 είναι πιο ανοιχτό για νέους συμμετέχοντες και δεν θεωρείται ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ μόνο για λίγου. Τώρα, κάποια άλλα σημεία. Και κλείνω με αυτά. Η ενδιάμεση αναθεώρηση, την είπε ο κύριο Σοντή. Κάθε προηγούμενο πρόγραμμα είχε μία ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, περισσότερο από ποτέ η ενδιάμεση ε, αναθεώρηση θα είναι πολύ σημαντική για τον ορίζοντα 2020, γιατί έτσι θα αλλάξει σημαντικά το κομμάτι αυτό και θέλουμε βεβαίω η ελκυστικότητα του ορίζοντα να συνεχίσει να υπάρχει. Ίσως βεβαίως αν χρειαστεί να λάβουμε και κάποια διορθωτικά μέτρα ως προς αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Οντί θέλει να πει κάτι. Πολύ πικρό, σύντομο. Εκφράστηκα άσχημα, εγώ ήμουν εισηγητής για την αναθεώρηση και είχα ρωτήσει μα μπορείτε να αλλάξετε τίποτα, μου είχαν πει αποκλείεται. Εγώ ζητώ μία αναθεώρηση των δημοσιονομικών προπτικών να αφήσουμε να ανασάνουν τα κράτη και μετά άμα θέλουμε εμείς 8 δις ε, για, ε, ε, το χρόνο να το απαιτήσουμε αυτό από το 2016 να αφήσουμε ήσυχα τα κράτη να κάνουν να, ανασάνουν στα, στα, στα, στους προϋπολογισμούς τους. Άμα δηλαδή πρόκειται να γίνουμε ρεζίλοι γιατί δεν θα τα βρούμε γύρω από τον προϋπολογισμό τώρα, ας αφήσουμε να πάρουν ανάσα μέχρι το 2016. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρία Ραμαδούρελη. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και την Κομισιόν και για τα σχόλια και για τη συνεισφορά τους. Εγώ τα σημείωσα όλα αυτά, διότι όλες αυτές οι συζητήσεις είναι πολύ χρήσιμες για να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Φάνηκε σαφώς ποια είναι τα σημεία που εκκρεμούν. Εγώ κατέγραψα έξι σημεία αλλά όλα αυτά είναι σημεία για, που, για, με τα οποία προχωρούμε, διότι θεωρούμε ουσιαστικό να έχουμε μία στεναρή θέση αυτού του Κοινοβουλίου. Εγώ θα σχολιάσω σύντομα μερικά ζητήματα. Εμείς μιλήσαμε πολύ για την ισορροπία του προγράμματος, τον, την ισορροπία 2020. Η κυρία Καρβάλιο το είπε καθαρά ε, και εγώ συμφωνώ, έχουμε ένα πρόγραμμα φιλόδοξο και καλοφτιαγμένο, γιατί ο βασικός μας στόχος είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί για να αναπτυχθούμε και να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό το σύστημά μας. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο σύστημά μας πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στην έρευνα και ανταγωνιστικοί στην καινοτομία. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί οι οργανισμοί, ε, οι ερευνητικοί μας οργανισμοί, τα πανεπιστήμια μας πρέπει να είναι ανταγωνιστικά θα πρέπει να διευρύνουμε την αριστεία, να έχουμε μια μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη της επιστήμης. Αυτό σημαίνει ισχυρό σύστημα. Πρέπει όμως να είναι και ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις μας, βελτιώνοντας τις τεχνολογίες τους που διευκολύνουν την καινοτομία. Να βελτιώσουμε την ιδιωτική χρηματοδότηση και να αυξήσουμε και τον αριθμό των καινοτόμων μήμη ε. Αυτό φαίνεται σαφές και στις τροπο, συμβιβαστικές τροπολογίες που συντάσσουμε τώρα, διότι ανησυχούμε για όλες αυτές τις πλευρές και προσπαθούμε να βρούμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ισορροπία. Είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό. Για τον προϋπολογισμό είναι μία από τις βασικές μας ανησυχίες, το ξέρουμε, φάνηκε από τη συζήτηση. Αλλά θέλω εγώ να ξεκαθαρίσω ένα θέμα. Η πρότασή μας είναι δική μας πρόταση και θα τσακωθούμε για αυτή την πρόταση μέχρι τέλους. Διότι πιστεύουμε στην πρότασή μας. Διότι εμείς έχουμε στοιχεία, έχουμε νούμερα, ξέρουμε τι έγινε με το τελευταίο πρόγραμμα πλαίσιο. <coughs> ξέρουμε το τι θα συμβεί στο μέλλον κάνει προβολές για το μέλλον. Ξέρουμε τι γίνεται με τους ανταγωνιστές μας, με την Κορέα, με την Κίνα, που επενδύουν σοριδών και αναπτύσσονται. Το Συμβούλιο θα κάνει την πρότασή του και ελπίζω να έχει εξίσου επιχειρήματα. Εγώ τώρα πιστεύω ότι πολύ καλά θα κάνουμε να συζητήσουμε, να συνεδριάζουμε και αν τα πράγματα δεν μας πάνε καλά, δεν θα υποχωρήσουμε. Θα ορίσουμε προτεραιότητες, αλλά θα τσακωθούμε όσο χρειάζεται, μέχρι τέλους. Και κάτι άλλο για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντήσω και να κάνω και δύο γενικά σχόλια. Ένα σχόλιο που εφαρμόζεται τόσο στην ασφάλεια όσο και στην ενέργεια. Εμείς μιλάμε για ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας. Δεν μιλάμε για πολιτικές ασφάλειας ή για πολιτικές ε, ενεργειακές. Μιλάμε για έρευνα και αυτό διευκρινίζει πολλά. Δεύτερον, η κυρία Γκουτιέρες Κορτίνες μας είπε το πώς θα οργανώνουμε, πώς θα εγγυθούμε τα μικρά σχέδια. Έχουμε διάφορες ε, τροπολογίες. Για τα flash flash play η συγγήτρια. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν τα σχέδια ναυαρχίδα. Συζητήσαμε επίσης το θέμα της διεύρυνσης της αριστείας και τα τμήματα τα οποία αφορούν στην τεχνολογία. Και σε όλα αυτά λοιπόν τα σημεία υπάρχει και υπάρχουν και τροπολογίες που αφορούν στα μικρά σχέδια. Εμείς είμαστε έτοιμοι σε όλες τις αλλαγές. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, θέλω απλώς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όλες τις υπηρεσίες αυτής τη επιτροπή, τα προσωπικά μας γραφεία που τέλος πάντων όλους όσους με τη βοήθειά τους μας βοηθούν στην η υλοποίηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Σημείωσα πολύ καλά και τις προτάσεις τους και τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Για κάποιες από τις παρατηρήσεις έχω και εγώ σχόλια να κάνω, αλλά σας λέω τα έχω σημειώσει όλα. Καταρχάς να τονίσω ότι το κριτήριο για την αριστεία του ορίζοντα 2020 είναι συμβατό με την διεύρυνση της συμμετοχής. Τι σημαίνει διεύρυνση της συμμετοχής? Σημαίνει ότι η αριστεία θα γίνεται σε μικρές μονάδες ε, που θα είναι διάσπαρτες ανά την Ευρώπη. Είτε είναι μικρομεσαίες, είτε είναι μικρές επενδυτικές, ε, ερευνητικές ομάδες, είτε είναι μικρά πανεπιστήμια. Όχι μόνο, δεν θα μιλούμε μόνο για μεγάλους παίκτες ή μεγάλα πανεπιστήμια ή μεγάλες βιομηχανίες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τα, τις, ε, τους όρους συμμετοχής με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορούν να συμμετέχουν και μικρές μονάδες που έχουν ε, τέτοιο επίπεδο αριστεία και θα μπορούν να υποφεληθούν από το πρόγραμμα. Το άλλο σημείο που ήθελα να δείξω είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα για την αριστεία. Τα διορθωτικά ταμεία είναι πρόγραμμα για δημιουργία ικανοτήτων. Έχουμε όμω δημιουργήσει κάποιε ενέργειε μεταξύ των δύο. Και έχουμε δημιουργήσει και αυτή την κλίμακα προ την αριστεία, το Stairway to Excellence. Και υπάρχουν συγκεκριμένε προτάσει. Έχουμε αναφέρει εδώ αρκετέ. Έχουμε κάποια αδερφοποίηση προγράμματα στα πλαίσια του, του ορίζοντα 2020 τα οποία βεβαίως μπορούν να διευρυνθούν, α πούμε για τη συμμετοχή περιφερειών που είναι απομακρυσμένε, που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα διαρθωτικά ταμεία. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά προγράμματα που υπάρχουν και μπορούν να συνδέσουν τα δύο αυτά προγράμματα η σφραγίδα της αριστείας που επίσης είναι, περιλαμβάνει κάποιες ε, σημαντικές προτάσεις αλλά δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τον ορίζοντα μπορεί όμως να χρηματοδοτηθεί από, τον, ε, από ε, τα διορθωτικά ταμεία αν η περιφέρεια από την οποία προέρχεται η πρόταση μπορεί να εμπίπτει στο, στα διορθωτικά ταμεία υπάρχουν λοιπόν πολλοί, πολλοί τρόποι για να, να συνδέσουμε τα δύο αυτά προγράμματα Επίσης, έχουμε μια ισόρροπη πρόταση κατά τη δική μου άποψη και προσπαθήσαμε να είναι όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη για την έρευνα και την καινοτομία καλύψαμε τον πλήρη κύκλο της καινοτομία και υπάρχει πάλι μία σύνδεση μεταξύ των διαφόρων κύκλων, γιατί υπάρχουν διαφορετικά, ε, διαφορετικές δέσμες προγραμμάτων. Νομίζουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ ισόρροπη πρόταση. Επίσης, για, τις μικρές, τις, για τα μικρά, μεσαία και μικρά προγράμματα. Έχουμε κάποια σχόλια που λένε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα μικρά ε, προγράμματα ε, και τα έχουμε συμπεριλάβει και αυτά στο ΦΕΣ και στις ε, προκλήσεις που υπάρχουν. Σε αρκετά σημεία λοιπόν του προγράμματος θα υπάρχουν μικρά project. Επίσης, η προστιθέμενη αξία της έρευνας. Η έρευνα είναι μία από τις πολιτικές όπου μπορούμε να δούμε ε, εμφανώς την ε, προστιθέμενη αξία. Η κριτική μάζα, η προώθηση της αριστείας, η αντιμετώπιση κάποιων πολύ σημαντικών ε, ε, προκλήσεων όπως ας πούμε οι σπανίες ασθένειες και η έρευνα πάνω στις σπανίες ασθένειες είναι το μίσο που μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα και σε ευρωπαϊκό και σε περιφερειακό επίπεδο. Και αυτό είναι, συμβαίνει και τα μεγαλύτερα ε, πανεπιστήμια της Ευρώπης Ας πούμε στη Βρετανία κάποια ε, πανεπιστήμια ε, έχουν υποφεληθεί από αυτό και είναι και σημαντικό το ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα πλαίσιο. Δεν είναι λοιπόν θέμα μόνο χρηματοδότησης. Σημαντικό επίσης είναι ότι υπάρχουν δίκτυα γνώσης που όντως καθιστά πολύ σημαντικό ε, να προωθηθεί αυτή η γνώση και για τις περιφέρειές τους αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης. Είναι λοιπόν σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την προσθέμενη αξία της ευρωπαϊκής έρευνας. Ευχαριστώ. Grazie alla collega Carvaio. Passiamo adesso al secondo Δεύτερο μπλοκ. Πέντε λεπτά ο συνάδελφος Έλερ. Θα σας κάνω πάλι να βαρεθείτε, ζητώ συγγνώμη. Ξεκινώ ίσως με το εξή. Στα πέντε λεπτά που έχουμε, μόνο κάποια επί της αρχής θέματα μπορούμε να αγγίξουμε Έχουμε πάνω από χίλιες τοπολογίες. Αλλά πιστεύω ότι για ένα τόσο περίπλοκο τεχνικού χαρακτήρα θέμα όπως τους κανόνες, κανονισμούς, rules, έχουμε υψηλό βαθμό συνένεσης. Ξεκινώ με την θεματολογική τοποθέτηση όπου υπάρχουν πολλοί συμβιβασμοί σε σχέση με την έκθεση αυτή που από πλευράς Ευρωπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή την αποδοχή των διεθνών μεθόδων λογιστικής από τους εμπλεκόμενους, απλουστευμένες διαδικασίες ε, ε, λογιστικών ελέγχων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εκτιμούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ε, εκτελεστικό συνέδριο, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να δομηθεί το σύστημα ελέγχων και λογιστικό σύστημα. Είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο δημοσιονομικό σύστημα που πρέπει να απλουστευτεί. Πρέπει να απλουστευτούν ολόκληρα συστήματα θεματολογικά και ίσως ε, όχι επί τρεις ή δύο ώρες με τους επαΐοντες θα πρέπει να συνέρθουμε, αλλά να μπορέσουμε σε, σε ε, σύντομο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για την απλούστευση. Και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως είχε, η δυνατότητα σε δύο βαθμίδες ε, τέτοιων λογιστικών ελέγχων και σε μία περίοδο έξι μηνών. Ξέρω ότι αυτό επιβαρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημιουργεί κάποια προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο εξαπλουστευτικό αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για, ε, πρέπει να απλουστεύει τα πράγματα για τους εμπλεκόμενους. Το θέμα της ελεύθερης πρόσβασης συνδέεται στενά με την, τον ορίζοντα 2020. Τεχνικά συνδέονται ε, ε, οι εκθέσεις ως προς αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή για μια ακριβή διατύπωση για το θέμα της ε, ε, ελεύθερης πρόσβασης νομίζω είναι σαφές ότι για τους ε, ερευνητές πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες και κανονισμοί που δεν θα δημιουργούν νομική αβεβαιότητα ή ανασφάλεια. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ της ελεύθερης πρόσβασης σε δημοσιεύματα και την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, τραπεζών δεδομένων ενώ η πρόσβαση σε, ελεύθερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν τίθεται να αμφιβόλο, έχουμε διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την ελεύθερη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή άλλα δεδομένα όπου πρέπει να διαφοροποιούμαστε. Τα πνευματικά δικαιώματα ε, παραγωγών, δηλαδή τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και η ελεύθερη πρόσβαση πρέπει να συνδεθούν μεταξύ τους. Συζητούμε αυτά τα θέματα αυτήν την εβδομάδα. Το όμως θα είναι υπέρ του ότι θέματα τα οποία είναι πολύ ευαίσθητα για το εμπόριο θα πρέπει να μπορούν να εξαιρούνται από τέτοιου κανονισμού και κανένα δεν πρέπει να υποχρεώνεται να δημοσιεύεται. Παρόλα αυτά ε, υποστηρίζουμε ω θέμα αρχή την κοινή προσέγγιση για την ελεύθερη πρόσβαση. Για το σύστημα αυτό τώρα των ποσοστώσεων ή των ε, αναλογιών, ένα, ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών είναι υπέρ της διασφάλισης ε, αυτή τη πτυχή ε, όσον αφορά τα πανεπιστήμια και την, ε, τους επιχειρηματικούς κύκλους και τις ε, βιομηχανίες όπως για την έκθεση Καρβάλιο, για την απλούστευση του πλαισίου είχε εγκριθεί. Πολλές τροπολογίες όμως χαρακτηρίζονται από πνεύμα συμπάθειας προς την απλούστευση που θέλει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με την επιστροφή των έμεσων δαπανών. Μια συζήτηση που δεν μπορεί όμως να ε, ξεχωριστεί απόλυτα από τα άμεσα κόστη. Υπάρχουν ε, ευρωβουλευτές που είναι υπέρ της πλήρους ε, κάλυψης του κόστους ή επιστροφής, όμως σε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμη μια τέτοια δυνατότητα. Στη διαφοροποίηση δεν είναι σαφές αν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, όσον αφορά τους ε, εμπλεκόμενους από τη βιομηχανία. Εάν αυτό θα ισχύει μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ΜΚΟ και πανεπιστήμια. Μία άλλη γραμμή είναι το θέμα των καταποκοπήν ποσών, flat rates, προτάσεις να αυξηθούν αυτά τα καταποκοπήν ποσά, προτάσεις μεταξύ 10% και 40% αύξησης σε σχέση με τα άμεσα κόστη. Το Συμβούλιο ήταν πιο μετριοπαθές σε σχέση με μια αύξηση από 20% σε 23% που συμφώνησε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τους σωστούς υπολογισμούς όλοι μας για να κατανοήσουμε περί τίνος πρόκειται. <clears throat> Δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε σχέση με τα κόστη ίσως ε, ε, τέτοιου είδους, ε, αποτελεσματικές τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Η δική μου πρώτη συμβαστική τροπολογία προσπαθεί αυτές τις τάσεις να τις ε, οδηγήσει σε σύγκληση. Πρώτον, με απλούστευση. Δεύτερον, με αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων. Και τρίτον, ε, δυνατότητα συγχρηματοδότησης. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ε, κάποιος αποκλεισμός ή κάποια ε, εξοδιαφοροποίηση όπως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο θέλουμε σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διατηρήσουμε την πρόταση αλλά να την συμπληρώσουμε όσον αφορά την πληρέστερη επιστροφή δαπανών που θα μπορεί ε, σε ένα συγκεκριμένο ύψος ε, να διασφαλίζεται. Αυτή είναι μια εναλλακτική λύση που προτείνεται. Δεν, να είναι, δεν θα είναι ε, υποχρεωτική. Όποιος θέλει θα συμμετέχει. Αν όμως επιλεγεί μια καταποκοπήν, ένας καταποκοπήν μια καταποκοπήν επιστροφή στον υπολογισμό, η συμβαστική πρόταση ε, επιτυγχάνει μια πιο δίκαιη επιστροφή για όσους συμμετέχουν στις ε, ε, δραστηριότητες έρευνας και που για παράδειγμα σε σχέση με τις κυριότερες ομάδες θα πρέπει να υποστηρίζονται. Πρέπει να έχουμε μια διαφοροποιημένη συζήτηση για αυτά τα σημεία. Θέλω να τονίσω, σημαντικό είναι να έχουμε close to market, να είμαστε κοντά στην αγορά και να δούμε τι γίνεται και με τα πανεπιστήμια. Έχουν μια άλλη δομή σε σχέση με την προσέγγιση στο close to market. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα της 100% κάλυψης ε, του κόστους ή των δαπανών. Την επόμενη εβδομάδα θα συζητήσουμε σε βάθος αυτά τα θέματα. Είμαι γνώμος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλή συνεργασία. Για όλα τα πρότυπα και προτάσεις από τους συναδέλφους ε, θα πρέπει να απεικονίζεται τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί σε σχέση με τα κονδύλια και ποιες επιπτώσεις θα έχουμε. Είναι μια σημαντική κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε, να δούμε ποια θα είναι η τελική έκβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκλάντε παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω μπορώ να αναφέρω τα εξής. Έχουμε βρει μια καλή μέθοδο θα έλεγα σε σχέση με τις τροπολογίες τις κατανείμαμε σε κατηγορίες. Υπήρχαν κάποιες κατηγορίες όπου βρισκόμαστε πιο κοντά ένας προς τον άλλον. Άλλα θέματα στα οποία πρέπει περισσότερο να συζητηθούν. Υπογραμμίζω το ότι για τα ποσοστά υποστήριξης έχουμε κάποια πρότυπα τα οποία είναι πιο απαιτητικά και φιλόδοξα σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα της, ε, του πλήρους υπολογισμού του κόστους ε, και της ε, επιστροφής ε, είναι σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν όλα αυτά. Σημαντικό είναι για μας ε, σε αυτό το σημείο, όχι όμως μόνο σε αυτό το σημείο, να βρούμε μια κατεύθυνση όπου υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα επιτυγχάνουμε κάτι παραπάνω και θα υποστηρίζουμε αυτές. Δεν πρέπει να είμαστε εχθρικοί προς τις ε, βιομηχανίες, αλλά οι βιομηχανίες μπορούν ε, και οι ίδιες α, αυτοτελώς να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υποστηριχθούν. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να δούμε τι θέλουμε ακριβώς να πετύχουμε και με ποιο κόστος και δαπάνες θα το πετύχουμε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να δημιουργούμε ολόκληρες δύσβατες περιοχές προσωπικών και άλλων δεδομένων που θα είναι πολύ δύσκολο να τις διαχειριστούμε και θα πρέπει να μην αφήσουμε να απολεστεί πρόσθετη αξία. Πρέπει να βρούμε μια σωστή αναλογία και σωστή ισορροπία των πραγμάτων. Δεν πρέπει να ανοίγουμε πόρτα και παράθυρο έναντι τρίτων χωρών να διευκολύνουμε αυτές τις χώρες σε σχέση με την προώθηση κάποιου προϊόντος τους, ε, με την δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας από πλευράς μας. Ε, θα πρέπει να είμαστε κάπως πιο σύνετοι. Και τελευταίο σημείο που πρέπει να συζητήσουμε είναι το κόστος διαχείρισης, οι δαπάνες διαχείρισης. Ε, μπορεί να είναι σκόπιμο να ανέρχονται σε ένα 7% ή σε ένα τέτοιο συγκρίσιμο πλαίσιο. Όμως πρέπει να δούμε αν πραγματικά είναι ανάγκη να γίνεται αυτό ή όχι. Πρέπει να προβληματιστούμε να δούμε μήπω το μέχρι σήμερα πρότυπο στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο μήπω θα ήταν πιο κατάλληλο. Και το κόστο το λογιστικό και το κόστο ε, των ε, υπολογισμών. Θα πρέπει να δούμε ότι από πλευρά κατών μελών έχουν γίνει σημαντικά βήματα πλούστευση ε, και η δυνατότητα συμμετοχή σε αυτό είναι σημαντική. Ευχαριστώ. Grazie. La collega Hall, prego. Κυρία Hall. Um, Ευχαριστώ. Και πάλι μιλώ εκ μέρους του κύριου Γιώχανσεν και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έλλερ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Για τον προπολογισμό ένα σχόλιο, γιατί ακούστηκε σε πολλές περιστάσεις. Ε, το πιο σημαντικό για το ΑΛΔΕ είναι να εξασφαλίσουμε ότι ο ορίζοντας 2020 θα παραμείνει στη θέση του, τη σχετική θέση που έχει μέσα στο πολιετέ ε, δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και στι διαπραγματεύσει που γίνονται. Γιατί έχουν ακουστεί τα, κάποια πράγματα ότι μπορεί ο προπολογισμό να πάει στο 40 δισεκατομμύρια, που είναι το μισό που έχει προτείνει η Κομισιόν και το μισό του 7ου προγράμματο πλαισίου. Γι' αυτό βεβαίω είναι τελείω απαράδεκτο. Ο κύριο Γιώχανσον λοιπόν θα ε, ήθελε να πιέσετε και εσείς και στις χώρες σας αλλά και εντός του Κοινοβουλίου για να μην φτάσουμε εκεί. Τώρα για την χρηματοδότηση. Υπάρχουν πολλές προτροπολογίες ε, για το μοντέλο χρηματοδότησης. Πριν όμως συμφωνήσουμε στη διάρθρωση του μοντέλου, αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι τι θέλει να επιτύχει αυτό το μοντέλο. Και στο Άλντε, Θεωρούμε ότι το εξή είναι σημαντικό. Ότι θα υπάρξει όντω απλούστευση για όποιου συμμετέχουν σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ότι το μοντέλο αυτό θα καθιστά πιο εύκολο ε, στα υπερεπιστήμια στου ερευνητέ τη ΜΜΕ να μπορούν να συμμετέχουν και ότι θα καταλήξει σε μια ε, ε, αυξημένη συμμετοχή της, του ιδιωτικού τομέα, τη βιομηχανία σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και επίση πρέπει να υπάρξει ευρεία συνένεση για τι λογιστικέ πρακτικέ που χρησιμοποιούνται από του διάφορου οργανισμού που χρησιμοποιούν αυτή τη χρηματοδότηση. Ακόμη και αν κάποιο έχει την καλύτερη ιδέα στον κόσμο, μπορεί να μην είναι πολύ έξυπνη αν αυτή η ιδέα τελικά οδηγεί σε περισσότερη γραφειοκρατία. Οπότε ίσως καλό θα ήταν να μην ε, εφεύρουμε κάτι από την αρχή, αλλά να προσπαθήσουμε να βασιστούμε στο σύστημα που υπάρχει και που χρησιμοποιούμε και που ξέρουμε ότι ε, λειτουργεί καλά σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμπερτς. Uh, uh, ε, τρία πράγματα για την έκθεση βεβαίως Βεβαίω, σα σημειώνω τα όσα είπατε πριν για τα στρατιωτικά. Εντάξει, το κατάλαβα αυτό που μου είπατε και χάρηκα που μου το είπατε. Λοιπόν, για το μοντέλο χρηματοδότηση. Αυτό που μας άρεσε στην πρώτη εκδοχή του Weller ήταν ότι όντως υπήρχε σαφώς διαχωρισμός, σαφής διαχωρισμός μεταξύ ερευνητικών ε, ε, ε, ιδρυμάτων, βιομηχανίας και πανεπιστημίων. Τώρα, είδαμε διάφορους πίνακες και τα διάφορα, από τα διάφορα μάλλον μοντέλα που προτείνονται και μας ανησυχούν κάποια από αυτά γιατί μπορεί να έχουν περίεργες συνέπειες εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Αυτό που θέλουμε είναι κάθε ε, λεπτό του ευρώ να αποτελέσει καταλήτη για την, για την ύπαρξη κι άλλων κονδυλίων. Είτε είναι από τον Ευρωπαϊκό Κορβανά, είτε μιλάμε για τις επενδύσεις των κυβερνήσεων, αλλά πέραν αυτού, κυρίως του, δικό του ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ε, ζωτική σημασία. Αν τώρα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου ουσιαστικά δεν έχουμε ε, ουσιαστική παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα με περισσότερα χρήματα, τότε κάνουμε λάθος κάπως στη δουλειά μας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οποιοδήποτε μοντέλο χρηματοδότησης διαλέξουμε, θα μεγιστοποιήσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Πιστεύω επίση ότι όταν μιλούμε για, την, ε, για το βιομηχανία, οι μικρότεροι παίχτε ουσιαστικά έχουν μεγαλύτερη ε, ανάγκη σε χρηματοδότηση από τι ε, από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μεγάλε επιχειρήσει μπορούν να αποτελέσουν τον καταλήτη για το πρόγραμμα, αλλά όχι για τη χρηματοδότηση, για τα κονδύλια. Και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα αυξήσουμε το μερίδιο αυτών. Ό,τι χρήματα δίνουμε στι εταιρείε θα πρέπει να αφορούν τι μικρομεσαίες εταιρείε κυρίω. Αυτή νομίζω θα πρέπει να είναι η βασική μα προτεραιότητα. Επίση, άκουσα τι είπατε για το fast track. Το fast track ε, δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το εργαλείο για, τα, για τις ΜΜΕ. Αν το fast track έρθει επιπλέον του ε, εργαλείου για τις ΜΜΕ, να το συζητήσουμε. Αλλά αν, το υποκαθιστά, δεν θα συμφωνήσω. Ε, για την ε, ανοιχτή πρόσβαση, όντω υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Η πρόσβαση στα δεδομένα θεωρούμε ότι είναι σημαντική. Και επίση πιστεύω ότι υπάρχουν ε, περιπτώσει, α πούμε, μια, για ένα project για το διαβήτη, όπου κάποια, ότι το MIT και η Novartis και το και κάποια πανεπιστήμια κάνουν προτάσεις για τον τομέα αυτό και διαθέτουν τα αποτελέσματα για τον, όλα τα δεδομένα ε, γιατί θεωρούν ότι θα βελτιώσει την καινοτομία. Ας δούμε λοιπόν και κάποια τέτοια παραδείγματα, ας δούμε που μπορούν να μας βγάλουν. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να συμφωνήσουμε, αλλά βεβαίως θέλουμε αυτή η συμφωνία να περιλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερους. Μη φοβάστε, όπως είπε και ο Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος. Η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να επιμείνω και να εμείνω στο θέμα το οποίο αναφέρθηκε για τη χρηματοδότηση και το οποίο έχει υποβληθεί ως πρόταση ε, συμβιβαστική. Ε, με κάποια ανησυχία αντιμετωπίζω αυτή την πρόταση για λόγους που προανέφερα. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει σαφής διαφοροποίηση μεταξύ πανεπιστημίων και ερευνητικών πανεπιστημιακών κέντρων και βιομηχανιών. Εντάξει, να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, παράλληλα σε σχέση με τις ε, ερευνητικές μονάδες. Αλλά υπάρχει και μεγαλύτερη δυσκολία σε σχέση με υψηλή έρευνα και που πιστεύω εγώ ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα την οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας. Απλούστευση, πολύ ωραία, εντάξει, αλλά Ποιο νόημα έχει η απλούστευση αν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα ή να ανταποκρίνεται αυτό το οποίο προτείνουμε στην πραγματικότητα. Και γι' αυτό έχω εδώ κάποια ανησυχία σε σχέση με την πρόταση για τα θεσμικά όργανα, για τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Θα πρέπει εδώ να δούμε τι γίνεται σε σχέση με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για να υπάρξει ενδιαφέρον που θα εκφραστεί από τα ερευνητικά κέντρα και σε σχέση και με την κάλυψη των ε, δαπανών εδώ πρέπει να δούμε και σε σχέση με την συμβαστική πρόταση. Κάποια θεσμικά όργανα δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Δεν θα έχουν το δυναμικό, δεν έχουν το δυναμικό να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία είναι όροι και προϋποθέσεις και που ζητούμε να ε, ακολουθούνται σε σχέση με αυτά τα κέντρα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τις ε, δυνατότητες επενδύσεων που υπάρχουν. Γι' αυτό πιστεύω εδώ ότι για το πρότυπο αυτό πρέπει να δούμε σε σχέση με τα θεσμικά όργανα και τα ε, ερευνητικά κέντρα για ένα ε, πρότυπο έρευνας για την ανάπτυξη, όμως δεν έχουμε δυναμικό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ε, απασχόληση για τους ερευνητές μας και τους νέους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε ότι πρέπει να υπάρξει έρευνα, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να απασχοληθούν μέσα στην έρευνα λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να καταβάλλονται οι αντίστοιχοι μισθοί και να είμαστε ε, στο επίπεδο εκείνο στο οποίο πρέπει να δράσουμε ε, ικανοί. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να προσλάβουμε νέους ε, ερευνητές και πώς θα μπορέσουν αυτοί να συνεργαστούν σε αυτά τα κέντρα τα ερευνητικά. Και πραγματικά με ανησυχία τα βλέπω όλα αυτά, διότι δεν πιστεύω ότι εδώ πρόκειται για μια καινοτομία, αλλά πρόκειται για μια αποκριστάλωση ενός συστήματος το οποίο δεν είναι το πιο ιδανικό θα πρέπει να δούμε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ένα πιο απλουστευμένο, ένα πιο λειτουργικό πρότυπο ώστε να μην υπάρχουν δυσκολίες και κίνδυνοι για τους ε, ερευνητές που θα θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν είναι δυνατόν ε, να αυτοϋπονομευόμαστε. Ευχαριστώ. Grazie. La parola alla collega per minuti, Anders prego. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής για τη σκληρή δουλειά πάνω σε αυτό το φάκελο. Το, ε, ο οργανισμός Ομπρέλα ε, που ουσιαστικά οργάνωσε την όλη αυτή, την, ε, όλη αυτή τη διαδικασία ε, την προηγούμενη εβδομάδα που συνεδρίασε συζήτησε τόσο πολύ το θέμα αυτό και δεν μπόρεσε να καταλήξει σε απόφαση για το αν θα, είναι, θα έχουν το καθεστώ του παρατηρητή. Η, η πολιτική για την καινοτομία δεν μπορεί να είναι πολιτική, είπε ο Γενικό Διευθυντή. Βλέπω όμω ότι τα μέλη εδώ τη ομάδα, της Επιτροπής σας δεν συμφωνούν. Θα ήθελα να μιλήσω τώρα για το θέμα της πρόσβασης στις περιπτώσεις όπου τα τεχνικά αποτελέσματα καλύπτονται από, τα, ε, ε, από τις πατέντες, από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, μπορεί να υπάρξει ένας κανόνας μη αποκλειστικότητας, όταν μιλούμε δηλαδή για αποτελέσματα δημόσιας χρηματοδότησης. Ε, ας πούμε, ε, κάποιες συνθήκες χωρίς ε, τέλη, αν ε, όμως διαγράψετε κάτι τέτοιο, ε, θα ήταν νομίζω ότι μεγάλο λάθος. Επίσης, για τη γενική απαγόρευση για το sub-licensing, όπως ε, είπε η Κομισιόν. Αν είμαστε σοβαροί για το τι θέλουμε να κάνουμε με την αγορά, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και τα μικρά project, χρειαζόμαστε όρου συμμετοχή που θα κινητοποιούν την καινοτομία και την έρευνα και θα έχουν και εφαρμοστε, εφαρμο, εφαρμόσιμους κανόνες, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε αποτελέσματα σε δεδομένα και αυτό προφανώ θα είναι πάρα πολύ αντιπαραγωγικό. Η ομάδα των Πρασίνων έχει υποβάλει κάποιε τροπολογίε που εξασφαλίζουν ότι θα υπάρχουν όλα αυτά, παρόλα αυτά αφήνουν και ένα περιθώριο ε, παρέμβαση ε, τη ε, της βιομηχανίας για ας πούμε μικρό χρονικό διάστημα, ότι πρέπει να, υπάρξουν μια, να υπάρξει μια καταληκτική ημερομηνία όπου η, θα πρέπει να εφαρμοστεί τελικά η ελεύθερη πρόσβαση. Για τι δημοσιεύσει και την πρόσβαση στις δημοσιεύσεις σε όλου αρέσει το πιλωτικό πρόγραμμα, σε όλα τα κράτη-μέλη, τέλο πάντων τα περισσότερα από αυτά έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση για την δημόσια έρευνα, κυρίω σε τέτοιε δημοσιεύσει. Για τα ερευνητικά δεδομένα, τα αποτελέσματα από τα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικά και προφανώ βοηθά το να βασίζεται στη, γνώμη, στη γνώση που υπάρχει ήδη από άλλου. Οι τροπολογίε των πρασίνων λαμβάνουν και αυτό υπόψη και εξασφαλίζουμε ευκαιρίε για, για τη διατήρηση των δεδομένων, έτσι ώστε να μην, ε, των, των άλλων δεδομένων, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να, ε, τρέξουμε σε, να προστρέξουμε σε ευαίσθητα δεδομένα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ή να χάσουμε με κάποιο τρόπο τα δεδομένα αυτά, γιατί προφανώς ε, δεν είναι σωστή αυτή η χρηματική διαχείριση. Οπότε έχετε το υπόψη σας. Ευχαριστώ, κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που με τέτοια προσπάθεια εργάστηκαν για αυτή την έκθεση. Πρώτα απ' όλα τον κύριο Έλερ που με εξαιρετικές προτάσεις και στη διαβούλευση τώρα για συμβιβασμούς προχωρούμε ώστε και στην Ευρωβουλή και αποκοινούμε το Συμβούλιο να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε στη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά. Τρεις παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Βρίσκω ότι αυτά τα οποία προτείνονται για πλούστευση και αναφέρονται σε σχέση με τους κανόνες για τη συμμετοχή είναι θετικά θα έλεγα για την κοινότητα των ερευνητών και για την ε, διάρκεια των έξι μηνών και για τα, τους λογιστικούς ελέγχους όλα αυτά βρίσκονται, είναι πολιτικές αποφάσεις ε, για τις οποίες από πλευράς Ευρωβουλής στο πολιτικό επίπεδο πρέπει να βοηθηθούν όσοι συμμετέχουν στην έρευνα. Δεύτερον, για την επιστροφή δαπανών, αυτή η διαφοροποίηση που γίνεται. Πρώτον, Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή γιατί για τους, τις διάφορες δραστηριότητες και τους υπολογισμούς διαφοροποιούνται τα πράγματα ανάλογα με τους ε, συμμετέχοντες και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται. Είναι σωστό αυτό και τα πανεπιστήμια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να υποστηριχθούν, να δούμε πώς μπορούμε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποστηριχθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε σε τέτοιου είδους επιστροφές ε, ε, δαπανών να λειτουργήσουν τα πράγματα σωστά. Και τρίτον, θέλουμε και οι βιομηχανίες να συμμετέχουν περισσότερο μέσα στον ορίζοντα, χρονορίζοντα 2020, περισσότερο από όσο συμμετείχαν υπό το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και αυτό πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας που πρέπει να είναι σεβαστά. Συμμερίζομαι την άποψή σας ότι πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά σε βάθος τι θα γίνεται σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τα αποτελέσματα των, ε, τα ερευνητικά, δημοσιεύσεις ε, κτλ. Πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα να μην ε, χάσουμε τα θετικά αποτελέσματα προσπαθώντας να ε, κάνουμε κάτι το ε, πιο σωστό. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε και η εμπορική εκμετάλλευση κάποιων θεμάτων να μπορεί και αυτή να καλύπτεται και να προάγεται. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τι παρεμβάσει όντω οι όροι τη συμμετοχή είναι πολύ σημαντικοί, είναι ο πυρήνα του προγράμματο πλαισίου. Τώρα, για τι ε, πρακτικέ ε, για, ε, για τα πρότυπα μάλλον τα λογιστικά. όντω υπάρχει τεράστια διαφορά στην Ευρώπη και θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Βεβαίω η αποδοχή αυτή α μην οδηγήσει σε κατάχρηση κάποιων πρακτικών. Αυτό πρέπει να το έχουμε επίση υπόψη για να μην δαπανίσουμε άσκοπα ευρωπαϊκά κονδύλια το εξάμεινο αυτό για τις επιδοτήσεις ε, πολύ φιλόδοξο. Ε, δεν νομίζω ότι θα το επιτύχουμε αν δεν έχουμε ε, ραγδαία πλούστευση των κανόνων. Είναι απλό το πράγμα. Και επίσης δεν θα πρέπει αυτό να ε, επηρεάσει αρνητικά το συνδυαζόμαστε να μπορούμε να οργανώνουμε αξιολογήσεις με πάνελ εμπειρογνωμόνων για να έχουμε και κάποιες απαντήσεις να δώσουμε σε όσους κάνουν αιτήσει. Τώρα, για την ανοιχτή πρόσβαση τα είπαμε και λίγο πιο πριν, υπάρχει το πιλωτικό πρόγραμμα. Ο κύριος Σέλλερ επίσης μίλησε για τη Rolls Royce. Αν η Rolls Royce όντως άφηνε, δημοσίευε τα δεδομένα που παίρνουν για, τα, για κάθε πρόγραμμα, τότε θα εξαφανιζόταν η η ανταγωνιστικότητα που έχει. Οπότε και αυτό θα πρέπει να το δούμε μάλλον προσεκτικά. Τώρα για το διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων ειδών συμμετεχόντων. Να σας θυμίσω ότι με τον ορίζοντα 2020 θέλουμε να ε, στηρίξουμε projects, όχι ε, συμμετέχοντες. Τα projects υπάρχουν για να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε κάποιους στόχους. Επίσης να σας θυμίσω ότι υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού Τρεις θα σας αναφέρω. Η συγχρηματοδότηση, ο, δηλαδή ο συμμετέχων πρέπει να συμβάλλει με κάποιο ποσό. Ε, η αρχή της, του μη κέρδου, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε κάποια ποσοστά που είναι ωφέλιμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Και ε, η ίση μεταχείριση μεταξύ των όσων θα συμμετάσχουν στα project αυτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. και επίση να μην ποινικοποιούμε τη βιομηχανία, γιατί η βιομηχανία είναι αυτή που θα πάρει την λαμπρή ιδέα και θα τη μετατρέψει σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα, προϊόν, διαδικασία και την αγορά και τελικά η βιομηχανία είναι αυτή που θα δημιουργήσει τις θέσει εργασία. Ούτε αυτό μην το ξεχνάμε. Τώρα, για τα έμεσα κόστη και τα flat rate, τα καταποκοπή ποσά, ε, από την εμπειρία μου σας λέω ότι τα έμεσα κόστη στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ήταν περίπου 30% του, λάθος που, ε, του ποσοστού λάθους που σημειώσαμε. Και ε, η ομορφιά της δικής μας πρότασης είναι, για να κάνω και λίγο διαβήμιση, ότι ε, για τα flat rates ουσιαστικά θα, θα καταρρύψει αυτό το 30% του λάθους, οπότε δεν θα χρειάζεται λογιστικός έλεγχος με το flat rate. Είναι σημαντικό λοιπόν και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Να σα θυμίσω επίσης ότι η εμπειρία δείχνει ότι οι συμμετέχοντες που έχουν πολύ ψηλά έμεσα έξοδα θα πρέπει μάλλον να δουλέψουν πολύ καλά ώστε να έχουν καλύτερο λογιστικό σύστημα γιατί ε, σημαίνει ότι έτσι μπορούν να ε, αλλάξουν τα έμεσα και τα άμεσα κόστη τους. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε προτείνει ένα συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμεσα κόστη. Και επίσης έχουμε και, τα, ε, και το κόστος διαχείρισης, που είναι ε, εν δυνάμει επιλέξιμο έμεσο κόστος. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει σωστή ισορροπία μεταξύ των ε, ισχυρών και των πιο μικρών, των πιο ευαίσθητων συμμετεχόντων, μικρών και μεγάλων εταιριών. Αυτό πρέπει να το δούμε πολύ λεπτομερώς, καθώς επίσης και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με το IPR, όταν έχουμε διεθνή συνεργασία. Ε, εκεί είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις δεν θα πρέπει να πηγαίνουν κατευθείαν σε άλλες χώρες χωρίς να αποφέρουν ε, ωφέλη και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής για να ολοκληρώσει. Συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα σας θερμά. Εδώ και δύο χρόνια σχεδόν περίπου το κάνουμε αυτό. Προπαρασκευή αυτών των δύο, αυτής της περίοδου δείχνει σε πιο υψηλό επίπεδο διεξάγονται οι συζητήσεις. Πεπειραμένοι συνάδελφοι όπως η κυρία Καρβάλιο που έκαναν αυτές τις προεργασίες και άλλοι, η κυρία Νίβλερ με πολυετή πείρα όταν εμπλέκονται σε αυτού του είδους τις συζητήσεις όχι επειδή εμείς θέλουμε κάτι νέο να επινοήσουμε, αλλά επειδή θέλουμε να έχουμε τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις που απαιτούνται, που είναι προϋπόθεση για ένα τέτοιο επιτυχές πρόγραμμα. Τις αρχές θα τις πω έτσι, ε, που πρέπει να σταθμιστούν και να αναλυθούν τις ανέφερα. Η μία είναι η απλούστευση, η simplification. Η άλλη είναι το leverage, η μόχλευση. Δηλαδή το θέμα ποιες άλλες επενδύσεις απαιτούνται στην έρευνα και καινοτομία και ποια είναι η μόχλευση που επιτυγχάνουμε. Η πορεία που καλύψαμε δείχνει ότι ενισχύουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη σκέψη της απλούστευσης με κάποιες προτάσεις που δεν είναι ιδεολειπτικές αλλά που βασίζονται σε κάποιους υπολογισμούς και που θα οδηγήσουν σε κάποιο συμβιβασμό που σίγουρα θα οδηγήσει σε απλούστευση αλλά από την άλλη πλευρά στη διαφοροποίηση αυτή θα διασφαλίζει για τους εμπλεκόμενους σε αυτά τα προγράμματα τη συμμετοχή τους σε αυτά ανάλογα με τις διαφορετικές τους ανάγκες πάντα. Διότι θέλουμε ένα πρόγραμμα ε, έρευνας και όχι να διευκολύνουμε απλά και μόνο χρηματοδότηση για οποιονδήποτε εμπλέκεται. Για το θέμα αυτό ανακουφίζομαι μετά από την παρέμβαση των πρασίνων συναδέλφων μας ε, με τις ε, προηγούμενες αντιπαραθέσεις που είχαν προϋπάρξει. Δεν πρόκειται εδώ σε σχέση με το 100% ε, πρόγραμμα κοινή ε, έρευνας. Έχουμε και στον τομέα των μεσαίων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στον τομέα των βιομηχανικών σημαντική συμμετοχή από επιχειρήσεις. Πρέπει να μεριμνήσουμε τα ε, συμφέροντα των πολιτών να μην υποστούν κάποια υπονόμευση σε σχέση για παράδειγμα με, τις, με τα διάφορα τηλεμετρικά δεδομένα που αφορούν για παράδειγμα κάποιες ε, ε, δράσεις π.χ. της ε, Rolls Royce ή άλλες. Ναι, θέλουμε ανοιχτή πρόσβαση. Θέλουμε και το σύστημα δημοσίευσεων στην Ευρώπη να συζητηθεί ανοιχτά. Και το θέμα της χρηματοδότησης βιβλιοθηκών, μητρών, αρχείων. Αν θέλουμε όμως ανάπτυξη, βρισκόμαστε σε ένα πεδίο ανταγωνιστικό, σε ένα πεδίο ανταγωνιστικών τάσεων και εντάσεων. Και εδώ πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε σε αυτόν τον ανταγωνισμό να είμαστε πιο ε, ανταγωνιστικοί και να είμαστε βιώσιμοι. Τελευταία παρατήρηση για το θέμα αρχής στον προϋπολογισμό για τα κονδύλια. Πρέπει να σκεφτούμε σε βάθος ότι ο προϋπολογισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε αναλογικότητα με τα διάφορα επιμέρους ε, στοιχεία. Τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί να γίνει με τα επιμέρους κονδύλια και ποια ποσοστά παρέμβασης μπορούν να προσφερθούν και να επιτευχθούν από πλευρά μα. Αν περικοπεί και μειωθεί ο προπολογισμό σε σχέση με τα κονδυλιά του, δεν θέλω να προδικάσω κάτι, αλλά το θέμα των ε, ουσιοδών σημείων δεν είναι ένα θέμα ε, συζήτηση σε ένα στεγανό. Πρέπει να διασφαλίσουμε επίπεδα παρέμβασης. Ο ίδιος προέρχομαι από την βιομηχανία, αλλά οι βιομηχανικοί κύκλοι έχουν ε, και την αρχή του καταλήτη ως ε, αρχική, ας το πω έτσι, αφετηρία και ως κυριότερο στόχο. Και θα πρέπει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι ιδιαίτερα καινοτόμες και αυτές να τις υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο τρίτο μπλοκ να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον κύριο Λάμπερτς. Madame uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρία πραγματάκια. Καταρχάς θα ευχαριστήσω, όλοι το κάνουν βέβαια, αλλά θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδες μου γιατί η συζήτηση νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επικοδομητική και αντικατοπτρίζει και τις ανταλλαγές απόψεων που κάναμε για τις υπόλοιπες εκθέσεις. Τρία βασικά σημεία ακανθόδη υπάρχουν ε, και έχουν μείνει έτσι για την έκθεση IT εκρεμή, πέραν του συνολικού προπολογισμού βεβαίως που είναι σημαντική συζήτηση τόσο ή άλλω ε, στην ε, όλη εξίσωση, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα σε αυτό. Καταρχά, η, επιλογή, η διαδικασία επιλογή. Ξέρετε, ως εισηγητής έχω προτείνει μια πολύ φιλελεύθερη φόρμουλα, ένα πολύ φιλελεύθερο τρόπο, ανταγωνιστικό, βασισμένο στην αγορά, όπου επιτρέπουμε το Συμβούλιο να επιλέξει εξάρτητο από τα ε, project που το επιβάλλονται, που του υποβάλλονται ανάλογα με την αξία που έχει το κάθε project. στα πλαίσια βεβαίω των θεματικών περιόδων που έχει το όλο ορίζοντα. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά έχετε εκφράσει ανησυχίε για το ότι θα πρέπει να υπάρχει και κάποιο βαθμό προβλεψιμότητα. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν έχει απασχοληθεί πάρα πολύ με το να προσπαθήσει να προβλέψει τον ρόλο της, ε, του Συμβουλίου και, της, και του Κοινοβουλίου για την ε, όλη διαδικασία επιλογής. Κάποιοι από τους ε, υποψηφίου μάλιστα διαφημίζονται και ω τέτοιοι. Ε, κατανοώ λοιπόν τις ανησυχίες σας. Ευχαριστώ να είμαι λιγότερο φιλελεύθερο από όσο ήμουν στην αρχή. Αυτό που δεν θέλω πάντως σίγουρα είναι να δώσουμε ένα, μια όθηση, ένα πριμ σε αυτούς που κάνουν πολύ καλό λόμπινγκ που ότι έχουν πούμε, λάβει μια α, επιβεβαίωση από την Κομισιόν ότι ναι, στο μέλλον θα σα προτιμήσουμε. Αυτό θα ήταν άδικο. Οπότε θέλω και αυτοί να πρέπει να τσουρουφιστούν λιγάκι όπω και οι υπόλοιποι. Ε, μπορούμε βεβαίω να μειώσουμε λίγο την ε, επιλογή μα σε ό,τι αφορά τι θεματικέ περιόδου, τι θεματικέ ενότητε που έχουμε έτσι ώστε να βρούμε μια ισορροπία. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να διατηρήσουμε ένα βαθμό ανταγωνισμού και ανοιχτού πνεύματος, γιατί αλλιώ δεν υπάρχει λόγος να έχουμε ε, ανεξάρτητο συμβούλιο ή Ένα λοιπόν είναι αυτό. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Δεύτερον, το θέμα της μόχλευσης πάλι. Επανέρχομαι με αυτό. Είναι γεγονό ότι το EIT είναι ο μόνο φορέας του, 20, ε, του ορίζοντα 2020 όπου είναι πραγματικά ε, ε, ε κομμάτι πυρήνα του γενικού προπολογισμού. Έχουμε 25 και 75%. 25 του ορίζοντα τα κονδύλια maximum 25 άλλα κονδύλια και το υπόλοιπο είναι ο ιδιωτικός τομέας ε, παρέμβαση και ίσως τα, υπερφερειακέ κυβερνήσει κυβερνήσεις ή ε, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Και θέλω να το διατηρήσουμε αυτό. Αν, αν ξεχάσουμε την, την ε, πτυχή της μόχλευσης, νομίζω ότι θα πάμε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που θέλουμε να πάμε. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε δυνατότητα παρέμβαση και είναι καλό να έχουμε δυνατότητα παρέμβασης. Ε, πρέπει αυτό να παραμείνει στην νομοθεσία. Και τέλο, η πρόταση αυτή ε, που έχετε κάνει κάποιοι για την περιφερειακή καινοτομία και τα διάφορα κονσόρτσια που υπάρχουν, έτσι ώστε να διαρθρωθεί αυτή η πολιτική, από κοινού με, τα, με την πολιτική και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ε, καλωσορίζω τι προτάσει αυτέ που έγιναν προ αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν βεβαίω κάποια στοιχεία που πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα συμφωνήσουμε. Πρώτον, υπάρχουν κονδύλια που να συνδέονται με αυτό και μπορεί να ακούγουμε λίγο κοινικό, κοινικός, αλλά αν δεν υπάρχει χρήμα γιατί νομοθετούμε. Ε, απλώς για να γράφουμε, αν δεν υπάρχουν πόροι. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και αν είναι έστω και μικρή αυτή η πόρη, έστω και λίγη. Αν δώσουμε κάποια χρήματα, ευχαρίστω να υπάρξει μια νομοθεσία. Αλλά δεν υπάρχουν ποσά, αν δεν υπάρχουν κονδύλια, τι νόημα έχει να το κάνουμε. Δεύτερον, Θέλουμε αυτά τα, αυτά τα κονσόρτσια να ε, συνδυάζονται με κάποια άλλα ή θέλουμε να να απευθύνονται κατευθείαν στο EIT. Εγώ θα προτιμούσα με κάποιο τρόπο τέλο πάντων να ε, συνδεθούν με κάποια από τα projects γιατί νομίζω ότι το EIT ε, ως βασική έτσι, δομή δεν κάνει ουσιαστικά δουλειά καινοτομίας απλώς οργανώνει τη δουλειά που κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν είναι το ίδιο. Νομίζω λοιπόν ότι για να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη αυτού του μέσου, καλό θα ήταν να το συνδέσουμε με τα υπόλοιπα. Και ε, κλείνοντας λέγω ότι υπάρχει και ένα θέμα, πώς να το θέσω, είναι κάτι έτσι ελεύθερο ή θέλουμε να επιλέξουμε κάποιους με βάση το δυναμικό της καινοτομίας που έχουν. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχει δυναμικό καινοτομίας ο υποψήφιος. Ακόμη και αν είναι μακροπρόθεσμο αυτό το δυναμικό. Πρέπει όμως να δούμε κάποιο δυναμικό. Γιατί αν ε, υπάρξει απλώς μια καλή δουλειά και δώσουμε και κάποιο μικρό κονδύλι, αλλά δεν υπάρχει δυναμικό καινοτομία, δεν βλέπω τι λόγο έχει υπάρξει σε αυτό το μέσο. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συνάδελφος Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω τώρα να πάω λίγο να, δω, τα δούμε αυτά. Ζητούν συγγνώμη σε σχέση με τους διερμηνείς για τις δυσκολίες ε, που ε, υπήρξαν πιο πριν. Θα ε, μιλήσω με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να αποσαφινιστούν τα δύο κυριότερα θέματα της έκθεσης για τους συμβιβασμούς που έχουν κατατεθεί και που έχουν συζητηθεί. Κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εισηγητές που συνεισέφεραν και υπέβαλαν τροπολογίες και προτάσεις για αυτή τη συζήτηση και που είναι καλοδεχούμενες αυτές οι προτάσεις. Θα επικεντρωθώ κυρίως σε δύο πτυχές. Η πρώτη αφορά ένα θέμα που ήδη αναφέρθηκε από τον συνάδελφο Λάμπερτ. Αφορά την ΚΙΚΣ, της κοινότητες αυτές ε, στην έρευνα. Είναι ένα από τα σημεία όπου υπήρχε η μεγαλύτερη διαφοροποίηση προτάσεων μεταξύ των προτάσεων των συναδέλφων. Και πρέπει να δούμε αν έχουμε όρους ε, για την, να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό υπό αυτούς τους όρους. Όπως εκφράστηκε από διάφορους συναδέφους από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, παρουσιάζεται ένας κλειστός κατάλογος, KICS, κλειστός κατάλογος μέχρι το 2020 και αυτό φαίνεται προβληματικό και σε μένα και σε άλλους που κατέθεσαν τροπολογίες. Αφενός είναι προβληματικό επειδή δείχνει ή φαίνεται ότι δείχνει ότι είναι η νίκη κάποιων λόμπις αυτή η κατάσταση που καταφέρνουν να κερδίσουν όσον αφορά το παιχνίδι αυτό το οποίο, στο οποίο, ε, το οποίο παίζουν ακόμα πριν ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Φαίνεται ότι αντιφάσκει αυτή η πρόταση σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέραμε για την αυτονομία της ε, έρευνας ε, ε, στο, στις δράσεις μας. Και δεν είναι αξιόπιστο να πούμε ότι στον τομέα της έρευνας με την καινοτομία πριν από συγκεκριμένες προθεσμίες θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε μέχρι το 2018 τα πιο σημαντικά πεδία. Και γι' αυτό η συγκεκριμένη αυτή ημερομηνία για το τρίτο κύμα ή την τρίτη ε, προσπάθεια, τρίτη κατηγοριοποίηση των ΚΙΚΣ και ιδιαίτερα όσον αφορά τις πολιτικές ε, της ε, πολιτικής, τις προτεραιότητες της πολιτικής και της έρευνας δεν μου φαίνεται ότι είναι το πιο εύθετο. Πρέπει να είναι ένα συμβιβασμός με όχι κλειστό κατάλογο αλλά μπορεί να αφήσουμε ανοιχτή την έκφραση των προτεραιοτήτων του Ευρωκοινοβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να υπολογίσουμε στον κανονισμό το θέμα της ε, παρουσίασης που πρέπει να είναι επαρκές ώστε νέοι υποψήφοι με νέες προτάσεις να μπορούν να συμπεριληφθούν. Να υπάρχει δυνατότητα για αυτούς τους νέους ανταγωνιζόμενους να βρεθούν σε ίσο πεδίο, σε ισότιμο επίπεδο με τους ανταγωνιστές. Ανταγωνιστές που όπως αναφέρθηκε ε, ποια είναι τα νέα θέματα των ΚΙΚΣ που ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είναι συγκεκριμένοι, επιλεγμένοι, εμπλεκόμενοι και πρέπει να μην αφήσουμε να είναι σε ένα κλειστό πλαίσιο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ε, έκφραση που ε, θα μπορεί να αφήνει σοβαρότητα στη δράση της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να αφήνουμε να ε, γίνεται κάτι το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει. Γι' αυτό πρέπει να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που θα εξισορροπεί την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θεμητά και νόμιμα, τις θεμητές και νόμιμες ανησυχίες των συναδέλφων και εμένα, ε, εμού της ίδιας επίσης. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω αφορά ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει αρκετές αντιφάσεις πρέπει στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε να πω ότι ε, το συζητήσαμε σε σχέση με την πρόταση για την έδρα του Ιδρύματος ε, Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Θα πρέπει στο συντομότερο ε, διάστημα να το αντιμετωπίσουμε. Σε σχέση με την έδρα στο Στρασβούργο που γνωρίζουμε ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να επιλύσουμε θέματα έδρας, για παράδειγμα, ε, αλλά όμως παρόλα αυτά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα της έδρας. Θα πρέπει να επιληθεί και να αντιμετωπιστεί έναντι των Ευρωπαίων πολιτών που πρέπει να τους δείξουμε τι κάνουμε με τα κονδύλια τους ε, όσον αφορά μια περίοδο λιτότητας ε, και που θέλουμε να δράσουμε αποτελεσματικά. Γι' αυτό αυτό που υπέβαλα είναι μια επικοδομητική θετική πρόταση που ε, σέβεται ιδιαίτερα την πόλη του Στρασβούργου που επελέγει ως έδρα και μέσα σε αυτή την θετική ε, τοποθέτηση θέλουμε να ζητήσουμε μία μελέτη, να συνταχθεί μία μελέτη. Μελέτη, Πρόεδρε, ο συμβιβασμό που προτείνω είναι η Επιτροπή από, πλευρά, από κοινού με το Συμβούλιο Διαχείριση ε, του Ιδρύματο θα υποβάλει μέχρι το 2015 τι ε, οικονομικέ λογιστικέ ε, πλευρέ και επιπτώσει για την ένταξη στην έδρα των κτηρίων του Στρασβούργου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των διευκολύνσεων στο Στρασβούργο τη έδρα αυτού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματο Τεχνολογία 2012, 2013, 2014, 15 και να μπορέσουμε με αυτή τη βάση να προχωρήσουμε και να μην υπονομεύεται το ότι θα μπορούσε να εξεταστεί αυτή η εναλλακτική λύση. Αυτά ήθελα να πω. Μια μελέτη να δούμε πώς θα μπορέσει αυτό να αντιμετωπιστεί για να διευθετηθεί αυτό το θέμα μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ματίας. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ να επενέστω την καλή συνεργασία που υπάρχει με όλους τους ανθρώπους για να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές προτάσεις σχετικά με το EIT. Στα περισσότερα θέματα έχει επιτευχθεί σημαντική προσέγγιση όπως επίσης σημειώνω και τα opinions που έχουν έρθει από άλλες επιτροπές που φαίνεται δείχνουν και σε αυτές τις επιτροπές να υπάρχει μια θετική εικόνα για το EIT. Έχουν μείνει δύο ανοιχτά θέματα. Ο κύριος Λάμπερτς και η κυρία Ματίας ήδη αναφέρθηκαν σε αυτά. Το ένα είναι πώς γίνεται η δημιουργία των νέων ΚΙΚΣ, πόσα και ποια θα είναι αυτά. Και εκεί προσπαθούμε όλοι με επικοδομητικό πνεύμα και με τις ανησυχίες που διατύπωσαν οι συνάδελφοι να βρούμε με ποιους τρόπους η διαδικασία των νέων ΚΙΚ θα μπορέσει να προσφέρει στη βιομηχανία, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα ένα ασφαλές και προβλέψιμο περιβάλλον για επενδύσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με αυτό που ο κύριος Λάμπερτς ε, ανέφερε, για αυτό που λέμε το τα δηλαδή το Regional Innovation Schemes, Ρώτησε ο κύριος Λάμπερτς αν υπάρχουν λεφτά. Φυσικά και υπάρχουν λεφτά, είναι το 5% του προϋπολογισμού του EIT, το οποίο προορίζεται για outreach και dissemination και συνεπώς μιλάμε για λεφτά. Φυσικά και είναι συνδεδεμένα με τα KICS, δεν θα είχαν άλλωστε καμία απολύτως έννοια εάν δεν ήταν συνδεδεμένα για το KICS και φυσικά μιλάμε για αριστεία και αυτός είναι ένας τρόπος, εάν κάθε ΚΙΚ μπορεί να έχει δύο-τρία τέτοια regional IS σχήματα πιστοποιημένης ε, ποιότητας, δηλαδή μένοντας κοντά στην excellence που θέλουμε, χωρίς να γίνεται ένας επιμερισμός απλώς ας δώσουμε και σε αυτή την περιοχή. Μένουμε στην αρχή της αριστείας είναι υπό την ομπρέλα των ΚΙΚΣ, αποτελούν τμήμα των ΚΙΚΣ και είναι ένας καλός τρόπος για να εμπλακούν οι τοπικοί πυρήνες αριστείας με τα ΚΙΚΣ που αποτελούν στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώ και είναι ένα καλό παράδειγμα από την Stairway to Excellence και πώς θα μπορούμε να κάνουμε προαγωγή αυτής της αρχής και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Τώρα για τρία λεπτά η κυρία Χόν παρακαλώ. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κύριο Λάμπερς για την πολύ καλή συνεργασία και την κυρία Ματία θα να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει για την επιλογή των ΚΙΚΣ θα ήθελα σε αυτό να αναφερθώ. Πολλές τροπολογίες έχουμε που αναφέρονται στην προσέγγιση 3 συν 3. Ε, εδώ θα πρέπει να το δούμε ξεχωριστά παρότι είμαστε φιλελεύθεροι, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει κάποια προβλεψιμότητα και κάποια βεβαιότητα, ώστε να ενδιαφερθούν οι επιχειρηματικοί κύκλοι και οι βιομηχανίες και να επενδύσουν και χρόνο και προσπάθειες για να ενταχθούν. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις όσον αφορά τα κίκς, αλλά και να διασφαλίζεται και κάποια ελαστικότητα. Εδώ θα υπαρκεστώ, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Είναι σαφής, σαφές ότι υπάρχει γενική συνένεση και υποστήριξη για τα ΚΙΚΣ. Το θέμα είναι στη διαφοροποίηση πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δεν λέμε τα ΚΙΚΣ δεν είναι σημαντικά καθόλου. Το θέμα είναι στη διαφοροποίηση, στις λεπτομέρειες όπως πάντα. Πώς θα διαμορφώσουμε τις λεπτομέρειες για να πετύχουμε το στόχο. Ευχαριστώ. Thank you uh, Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους <clears throat> Δεν είμαι σκιώδη εισηγήτρια, θα ήθελα όμω να γνωμοδοτήσω κι εγώ, μια και σε μεγάλο βαθμό εμπλεκόμουν σε ε, κάποια από αυτά τα θέματα. Πρώτον, το αποτέλεσμα μόχλευσης και σε σχέση με τα κονδύλια των διαθετικών ταμείων, τι μπορεί να γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, να δούμε ότι αυτό είναι επίση ένα τρόπο να μπορέσουν να διευρυνθούν οι δυνατότητε από πλευρά ε, κονδυλίων οι δυνατότητε τη έρευνα και καινοτομία, όχι μόνο με το τον ορίζοντα 2020, αλλά και τα ποσοστά και των κονδυλίων των ε, Διεθνικών ταμείων που θα αφιερωθούν σε αυτούς τους στόχους. Συμπληρωματικά, να μην υπάρχει επικάλυψη, αλλά να προηλυένεται το έδαφος και να προετοιμάζονται όλα αυτά α, κατάντι και ανάντι, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση με καινοτόμο τρόπο να διασυνδέσουμε όλα αυτά και τα κίξ όχι μόνο στις κυριότερες, ε, στα κυριότερα δομικά του στοιχεία αλλά στην αναβαθμισμένη ποιότητα που πρέπει να επιτευχθεί σε σχέση με τα κίξ να μπορέσουν ε, να επιτευχθούν ε, αυτές οι ομαδοποιήσεις και αυτές οι στοχοποιήσεις να μπορέσουν να εμπλακούν με αυτόν τον τρόπο στην δημιουργία πρόσθετης αξίας και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τα ε, διαθροτικά κονδύλια και τη μόχλευση και από τα διαθροτικά ε, ταμεία και κονδύλια. Θα πρέπει να ε, πούμε ότι ο κυριότερος όγκος δεν είναι ο όγκος των ΚΙΚΣ, είναι μια διαφοροποίηση που εδώ πρέπει να γίνει σε σχέση με τις χρήσεις, με ιδιαίτερα προσεκτικό τρόπο, για την επιλογή και επιλεξιμότητα. Συμφωνώ απόλυτα σε σχέση με την διατύπωση της Fiona Hall. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι σε σχέση με τις δυνατότητες προσέλκυσης ε, των βιομηχανιών και κάποιου βαθμού ε, ευελιξίας. Το τελευταίο σημείο, το χρονοπλαίσιο για την ανάπτυξη και εξέλιξη αυτού του σχεδίου. Πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη χρονική ε, διάρκεια διότι θα πρέπει να δούμε και ένα μεγαλύτερο χρονορίζοντα για την συμμετοχή των όσων θα εμπλέκονται πέρα από το τριετές πλαίσιο ε, που ε, προβλέπεται. Ευχαριστώ. ich möchte noch mal einen äh, Θα ήθελα για μια στιγμή να δώσω κάποια διαφοροποίηση στην τοποθέτησή μου είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο αυτό. Ωστόσο πρέπει να το συγκρίνουμε με το επίπεδο αξιολόγησης που, του οποίου έτυχαν άλλα προγράμματα ε, στο παρελθόν και γνωρίζουμε για το EIT σχετικά λίγα πράγματα μέχρι σήμερα. Ε, έγιναν κάποια πράγματα σε μια χρονική στιγμή όπου τα ΚΙΚΣ σε μεγάλο βαθμό δεν είχαν καν θεσμοθετηθεί και δεν λειτουργούσαν και έχουμε μια, ένα δεκαπλασιασμό των κονδυλίων όσον αφορά τη μόχλευση. Αν λάβουμε υπόψη τις φιλόδοξες ε, δομές για τη συγχρηματοδότηση ή χρησιμοποιήσουμε αυτές ως βάση, τι θα σημαίνουν όλα αυτά. Η βιομηχανία με έναν παράγοντα στην ιωστή δύναμη ή στην δύναμη Χ θα πρέπει να είναι πρόθυμη να προβεί σε επενδύσεις για να είμαστε αποτελεσματικοί. Να εκφράσω εδώ το τι σημαίνουν όλα αυτά. Δεν έχουμε κάποιες εμπειρικές ε, εκ των τεκμηρίων ε, προοπτικές ότι όλα αυτά θα μπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν σε μια πρώιμη φάση αυτού του προγράμματος. Απλό ερώτημα, μήπως το ίδιο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με πολυτεχνία ή τεχνικά, τεχνικές ανώτατες σχολές στα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα και πρέπει να απαντηθεί. Γι' αυτό θέλω κάποιες επιφυλάξεις να εκφράσω εδώ από πλευρά μου, διότι δεκαπλασιασμός των κονδυλίων σε μια τόσο πρώιμη φάση αυτού του σχεδίου, χωρίς μια σε βάθος αξιολόγηση αυτού του προγράμματος, αυτού του σχεδίου, ή είναι κάτι το εξαιρετικά φιλόδοξο, δεν θέλω να το αποκλείσω αυτό, ή βασίζεται σε κάποια στοιχεία που δεν είναι τα αναγκαία στοιχεία αξιολόγησης, όπως εκείνα τα οποία λαμβάνουμε υπόψη πάντα σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις όταν αξιολογούμε ένα άλλο πρόγραμμα ή σχέδιο. Αυτό πρέπει να λάβουμε υπόψη. Τώρα για το ERC, με ποιο τρόπο ε, σταθμίστηκαν τα πράγματα ή αξιολογήθηκαν. Ε, όλα αυτά δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά τα οποία κάνουμε τώρα με τα EIT. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Ο κύριος Οντί, δύο λεπτά παρακαλώ. Πολύ σύντομα για την έκθεση Λάμπερτς. Εγώ αναρωτιέμαι για το ρόλο της, ε, του Ιδρύματος. Εμείς έχουμε, ε, το λέω ως εισηγητής δηλαδή, ε, στη, για, για, την ε, αξιολόγηση του προγράμματος, έχω προβλήματα, έχω αμφιβολίες. Δείτε εμεί τι επίδραση έχουμε με όλους όλους αυτούς διευθυντές, υπαλλήλους, διοικητικά συμβούλια και τα λοιπά των διαφόρων οργανισμών. Όλα αυτά τα διοικητικά συμβούλια δεν καταφέρνουμε να τα ελέγξουμε. Ακόμη και όταν έχουμε αρνητικές ε, απαλλαγές προϋπολογισμού, δεν ξέρουμε, γιατί είμαι και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, δεν ξέρουμε ποιε θα είναι οι κυρώσει που παίρνονται, διότι έχουν την, από τα διοικητικά συμβούλια που είναι αυτόνομα. Και πρέπει πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ανάκλησης των ε, ε, των διοικητικών συμβουλίων ε, και οι προσλήψεις πρέπει να γίνονταν ανεξάρτητα και για την έδρα του Κοινοβουλίου είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι εδώ, δεν είναι θέμα να το συζητήσουμε εδώ, αλλά δεν είναι και καν θέμα του ντοσιέ αυτού. Η Κομισιόν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ στον εισηγητή και, και το σκεώδη εισηγητή. Εγώ πιστεύω ότι μετά που έγινε η πρόταση της Κομισιόν ε, ορίζοντας 2020 έχουμε κάνει μεγάλες πρόοδους και μας επέτρεψε και στην ΙΤΕ και στους ΚΙΚΣ να παρουσιάσουμε σωστά ό,τι έγινε μέχρι τώρα μας επέτρεψε να έχουμε μία συζήτηση πιο ήρεμη, εστιαζόμενη ε, στα πραγματικά προβλήματα. Τώρα, πρώτο σημείο. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Έλερ για τα ΙΤΕ και τα ΚΙΚΣ, που μας λέει ότι είναι καινούρια ε, εφευρήματα και δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε τώρα. Γι' αυτό η Κομισιόν είπε δύο φάσεις. Μέχρι το 2018 μία πρώτη φάση και όταν έχουμε αναθεώρηση το 2018 και είναι θετική η αναθεώρηση τότε να απολευθερώσουμε και, τη δεύτερη, και το δεύτερο τμήμα του στον προπολογισμό. Μετά τα τρία σημεία τα οποία ανέφεραν οι δύο συνεισηγητές, ο κύριος Λάμπερτ και η κυρία Ματίας και τους ευχαριστώ για το πόσο αναλυτική ήταν το θέμα για την επιλογή των ΚΙΚΣ. Ε, θεωρούμε ότι αυτό συνδέεται με την ίδια τη φύση του ΚΙΚ. Το ΚΙΚ για να είναι πραγματικά ΚΙΚ και για να είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουμε στα πλαίσια της έρευνας ή του ορίζοντα 2020 πρέπει να είναι ένα διαφορετικό ζωάκι, μια κάτι διαφορετικό. Πρέπει να ε, βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο της γνώσης και να έχει και τη δυνατότητα χρηματοδότησης ε, και αηφορίας. Γι' αυτό λοιπόν τα κίξ είναι διαφορετικά. Δεν πρέπει εμείς να έχουμε ένα σωρό κίξ τα οποία δεν θα είναι κίκ αλλά θα είναι διαφορετικά πράγματα. Θέλω λοιπόν να κάνω δύο διευκρινήσεις. Κατά την τωρινή περίοδο στον κανονισμό κίκ που ισχύει σήμερα τα θέματα τα αποφασίζει ο νομοθέτης, δηλαδή Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Στα πλαίσια τροποποίησης ε, του κανονισμού ΙΤΕ, η Κομισιόν και απόλυτα συνεπής με την κατάσταση, πρότεινε να γίνει συζήτηση για τη θεματολογία και βάση κριτηρίων. Σας δώσαμε προτάσεις ε, με κριτήρια σαφή, μετά από δημόσια διαβούλευση, αλλά να σας πω σαφέστατα ότι επειδή ήδη η Κομισιόν η Κομισιόν με τρόπο ιδιαίτερα ανοιχτό και διαφανή αποφάσισε θέματα. Θέματα τα οποία εμπνέονται από τον ορίζοντα 2020. Και ο νομοθέτης λέει ότι αν δεν είναι αυτά τα, τα θέματα που ενδιαφέρουν τότε να τα αλλάξουμε. Αλλά μη μας λέτε ότι έχει προδικάσει ήδη τη θεματολογία ή η Κομισιόν. Λοιπόν, δεύτερο σημείο. Τα, τα ΙΤΕ, ή 25, 75 κλπ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τα ΚΙΚ φτάνουνε. Αν προσθέσουμε όμως και άλλες δεσμεύσεις και αν κωδικοποιήσουμε ε, και αν ορίσουμε με υπερβολική ακρίβεια από πού έρχονται τα άλλα ε, κονδύλια, τότε πραγματικά κινδυνεύουμε να δολοφονήσουμε το ζώο, λέει ο μιλητής. Πρέπει να, να το, το 2575 χωρίς να πούμε τίποτα παραπάνω. Ο κύριος Τσουκαλάς μας θύμισε ότι ήδη υπάρχει μία πρόταση που λέει ότι το 5% θα πρέπει, του προπολογισμού πρέπει να πηγαίνει σε αυτές τις δραστηριότητες. Λοιπόν, και βεβαίως κύριε Λαμπέρ, εμείς μπορούμε κάλλιστα να νομοθετήσουμε για ένα προπολογισμό. Ε, βάλτε μία πρόταση στο τραπέζι. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε την δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας αυτές ε, μπορούν να έχουν νόημα όταν εντάσσονται μέσα στη γενικότερη προσπάθεια όπως είναι τα κίτσια, διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος διάχυσης. Ο κύριος Λάμπερτς. Να απαντήσω. Θα ξεκινήσω μετά ως όσα Μπορώ να σας πω ότι για το για τα... Υπάρχουν εκεί που έχουν, μάλλον υπάρχουν κάποια κονσόρτσια που ε, ακόμη και στο ίντερνετ διαφημίζονται ότι ήδη έχουν επιλεγεί. Ίσως να έχουν παραερμηνεύσει αυτά που τους είπατε, αλλά υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι που ε, ήδη θεωρούν ότι είναι, έχουν επιλεγεί. Ο στόχος ενός κικ είναι να μπορεί να λειτουργήσει μόνο του τελικά. Οπότε για μένα μπορεί να είναι ανοιχτό το περιθώριο. Βεβαίω είναι λογικό, σε τακτική βάση θα αξιολογούμε αν έχει υπάρξει πρόοδο. Αν δεν υπάρχει στενή εποπτεία, μάλλον αν υπάρχει στενή ε, εποπτεία χωρί όμω οικονομικέ συνέπειε, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τεράστια πειθαρχία. Τα έχουμε δει και στην οικονομική διακυβέρνηση αυτά. Χρειάζεται δηλαδή πραγματική παρακολούθηση. Και κάποια ορόσημα που θα μας επιτρέψουν να δούμε πόσα χρήματα θα δίνουμε και για πόσο χρόνο. Αν θέλουμε κάποια πειθαρχία πρέπει να είμαστε αυστηροί. Για την αξιολόγηση. Κρίστιαν, συμφωνώ μαζί σου. Το να δίνουμε έτσι κονδύλια σε κάτι που δεν αξιολογείται δεν είναι σωστή χρηστή διαχείριση. Αλλά για, με τα JTI τι γίνεται. Το EIT δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ένα JTI και δεν ξέρω αν έχουμε και πολύ καλή αξιολόγηση για τα JTIs. Αν έχουμε αξιολόγηση καταρχάς. Και αυτό δεν σημαίνει ότι, δεν κάνουμε, ότι αν κάνουμε κάπου κακή διαχείριση πρέπει να κάνουμε και κάπου αλλού κακή διαχείριση. Όχι. Αλλά α μην είμαστε βασιλικότεροι του βασιλέω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ισόρροπη προσέγγιση. Κατανοώ αυτό που λες, αλλά από ό,τι βλέπω εγώ και από τι απαντήσει που έχω λάβει, πολλοί εμπλεκόμενοι φορεί λένε ότι πάει στην καλή κατεύθυνση το ζήτημα αυτό και δεν έχει μείνει ανεξέλεγκτο. Δεν λέμε πάρτε τα δισεκατομμύρια και κάντε τα ό,τι καταλαβαίνετε και σε 7 χρόνια θα τα ξαναπούμε. Δεν προτείνουμε αυτό πάλι θα έρθω στο θέμα τη εποπτεία. Εγώ είπα να, κάνουμε, να κάνει το Κοινοβούλιο ετήσια αξιολόγηση του τι γίνεται. Ίσως στο κάθε EIT θα πρέπει ίσως να, να ε, ε, εξελιχθεί σε, για όλο το πρόγραμμα, όπως κάναμε με τον Τράγκη, που τον βλέπαμε κάθε τρει μήνες. Δεν ζητώ κάτι τόσο αυστηρό, αλλά για να απαντήσω και στο Σαμπιέρ ce que je veux dire c'est qu'on euh, peut, aussi exercer notre rôle de contrôle θα μπορούσαμε λοιπόν να ελέγχουμε, να κάνουμε, εξασκήσουμε το δικό μας ρόλο του ελέγχου, έτσι ώστε να μπορεί και η κάθε, να μπορούμε να ζητήσουμε από, την κάθε, από το κάθε εμπλεκόμενο φορέα να έρθει και να δώσει εξηγήσει. Αν αυτό χρειάζεται βεβαίω. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε απλώς τα ιδιωτικά κονδύλια. Δεν είχα την ευκαιρία να το συζητήσω με τους συναδέλφους, αλλά θα, το, θα συνεχίσω κι εγώ να το παρακολουθώ. Σενιόρα Ματίας, τρεις μινούτους. Κυρία Ματίας, τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για τα σχόλια που έγιναν. Επίσης, θα απαντήσω μόνο σε κάποια από τα θέματα που αναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αποσαφηνήσω ότι ποτέ δεν είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποκλείσει ποιοι θα έπρεπε να εμπλέκονται, εκείνους που θα ε, εντασσόντουσαν στα ΚΙΚΣ. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε ήταν το ότι υπάρχουν δυνάμει συμμετέχοντες που αναφέρονται ως μελλοντικοί συμμετέχοντες της, ε, των ΚΙΚΣ. Αυτό είναι διαφορετικό. Δεν ετίθετο αυτό με κανένα τρόπο ε, ε, ε, εις βάρος της Επιτροπής. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα ε, πρότυπο το οποίο θα μπορεί να συνδυάζει την ικανότητα σε μια ανοιχτή δυνατότητα επιλογών και θα δίνει ισότιμο πλαίσιο συμμετοχής σε όλους που θα εμπλέκονται στα θέματα που συνδέονται με τον ορίζοντα 2020. Δεν κάνουμε λόγο για άλλο πράγμα παρά μόνο γι' αυτό. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα και δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Λοιπόν, διατηρώ αυτό, παραμένω σε αυτά τα οποία είπα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το, χέρι, από το χέρι μας να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Και για τα θέματα του EIT, του Ιδρύματος Τεχνολογίας ε, και Καινοτομίας, με τα όσα προτάθηκαν, θα πρέπει να είναι ένα καλό πρότυπο, ένα καλό, μια καλή δομή σε σχέση με τις ε, δυνατότητες που θα μας παρέχονται. Δεν έχουμε άλλα δυνατότητα, δεν μπορεί να υποκατασταθεί ή να συγκρίνεται με το ρόλο των τεχνικών πανεπιστημίων ή των πολυτεχνείων. Δεν είναι συγκρίσιμο. Το μόνο μέσο που έχουμε και που αναφέρθηκε πολλές φορές είναι η παιδεία, η έρευνα, η βιομηχανία, η ε, έρευνα μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Και πρέπει εδώ να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε πρόσθετη αξία από τις δράσεις μας, σε μεγαλύτερη δημιουργία απασχόλησης και μεγαλύτερες επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Αυτά είναι πρόδειλα, είναι προφανή ότι έτσι πρέπει να διαμορφωθούν και να υπάρξει και αξιολόγηση και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε είναι προφανές ε, ότι θα πρέπει να δοθούν ε, τα εχέγγυα ώστε να υπερψηφιστεί αυτό το πρότυπο και να διασφαλιστούν τα κονδύλια από πλευράς προϋπολογισμού. Τούτων λεχθέντων και για να ολοκληρώσω και μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, Πρόεδρε, ολοκληρώνω, ολοκληρώνω λέγοντας, συνάδελφε οτί λέτε ότι μπορούμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία σε αυτό το θέμα. Να δούμε και το θέμα της έδρας ε, του στο Στρασβούργο για το Ίδρυμα ε, Τεχνολογικής ε, Ανάπτυξης και Έρευνας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πώς θα μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το όργανο και πρέπει πραγματικά να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο ένα θέμα της ε, γαλλική κυβέρνησης της Γαλλίας ή της πόλης του Στρασβούργου. Είμαστε όλοι μας εδώ εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και πρέπει να προχωρήσουμε να βρούμε μια λύση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Συγγνώμη κυρία Ματία, νόμιζα ότι ε, ήταν δύο τα λεπτά αλλά ήταν τρία. Εντάξει, ολοκληρώσατε. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που αναφέρεται στο πρόγραμμα έρευνας και κατάτησης της Ευρατόμ. Και θα λάβει τον λόγο για πέντε λεπτά ο κύριος Σκίνερ, παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ. Θα χαρείτε, γιατί δεν θα μιλήσω για όλο το χρόνο που μου έδωσε ο Πρόεδρος, κυρίως γιατί έχουμε μεγάλο βαθμό συμφωνίας όπως είπα και την προηγούμενη φορά, όταν μίλησα στην Επιτροπή, ε, υπήρχαν αρκετές τροπολογίες οι οποίες υποβλήθηκαν. Κάποιες ε, τις, ε, μπόρεσα να τις συμπεριλάβω, οπότε βελτιώθηκε το κείμενο. Ευχαριστώ όσους τις υπέβαλαν. Και με την ευρία αυτή συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει και στι ομάδε και στην Επιτροπή, σίγουρα θα έχουμε ισχυρή φωνή ω Κοινοβούλιο στο θέμα αυτό και απέναντι στην Κομισιόν και εκτό. Δύο ε, συμβαστικές προτάσεις έχω υποβάλει σε ό,τι αφορά το, την χρηματοδότηση. Έχουμε μια συνεκτική γραμμή, ε, όπως αυτή που μας πρότειναν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Προϋπολογισμού, έτσι ώστε να έχουμε μια, ε, ένα σαφές, έναν σαφή τρόπο και διαφανή για την χρηματοδότηση. Ελπίζω να, μπορεί, να μπορούν και οι υπόλοιπε ομάδες και οι σκιώδες να τις συζητήσουν πέραν των όσων έχουμε ήδη συζητήσει. Ξέρω ότι ήδη συζητήσαμε κάποια, κάποια πράγματα πριν έρθω εγώ εδώ ε, Βιτόριο, εσύ ανέφερε ε, κάτι για το α, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, Βεβαίω δεν περιμέναμε να είναι έτσι ε, εκ πρώτη όψεω το πράγμα, αλλά πρέπει να περιμένουμε ότι στα πλαίσια και στο ανώτατο όριο που θα έχει το MFF θα μπορέσουμε να το περάσουμε. Ε, ήμουν εδώ την προηγούμενη Πέμπτη όταν γινόταν μια συζήτηση με τον ε, Επίτροπο Έτινγκερ και ήρθε, όπου ήρθε να μας παρουσιάσει, του, ήρθε μάλλον στο, στη συνάντηση των ε, συντονιστών για να σχολιάσει τα stress tests ε, με τα οποία είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά η έκθεσή μου συνεχίζει να τονίζει ότι δεν έχει να κάνει με το stress test, αλλά υπάρχει ένα, μια πτυχή που τονίζει ακριβώς την ειδική ανάγκη για κατάρτιση και για ασφάλεια στον τομέα αυτό. Γιατί αν πρόκειται να έχουμε μια ε, ασφαλή πυρηνική βιομηχανία, πρέπει η ασφάλεια να μπει ως ε, προαπαιτούμενο ε, στις συζητήσεις που θα κάνουμε με τους επιστήμονες στην, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχουμε πει μέσω των διαφόρων τροπολογιών ότι αυτό θα είναι ένας από τους τομέας όπου θα πιέσουμε πολύ. Ε, αν ας πούμε το decommissioning ήταν ε, ένας από τους σημαντικούς φορείς, θα πρέπει ε, να αποτελέσει συγκεκριμένη πτυχή και για την κατάρτιση και για τους επιστήμονες που θέλουν να το παρακολουθήσουν σε επίπεδο πανεπιστημιακό, ακαδημαϊκό. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν δούμε τον υπόλοιπο κόσμο, πρέπει και εμείς να είμαστε σίγουροι ότι αν δεν υπήρχαν οι Ευρωπαίοι επιστήμονες, θα έπρεπε να βασιστούμε όχι στους καλύτερους ε, του κόσμου. Ελπίζουμε όμως ότι εμείς θα είμαστε μέσα στους καλύτερους αυτού του κόσμου με αυτά τα project. Δεν νομίζω ότι ε, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Με αυτά λοιπόν, α, ε, Πρόεδρε, εγώ θα σταματήσω εδώ και ελπίζω να μπορούμε να συνεχίσουμε. Relax. Πάντοτε θα έχετε τη συνένεσή μου. Η κυρία Ριβαζή. Για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε η πράσινη είναι κατά και επί της ουσίας και επί της μορφής της συνθήκης ουρατόμα. Διότι πρόκειται ε, για τη ενθάρρυνση της πυρηνικής ενέργειας που είναι πια ξεπερασμένη επί της ουσίας και επί ε, του τυπικού διότι δεν τηρείται η συναπόφαση. Εμείς εδώ πάντοτε παλεύουμε για τη διαφάνεια. Και για τα πυρηνικά το βασικό είναι να μην έχουμε συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών. Ο κύριος Σκίνερ μας μίλησε για την παρέμβαση του κυρίου Έρτιγκερ για τα stress test. Και επ' αυτού οι πολίτες ζητούν απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τα stress test πράγμα το οποίο ναι μεν ε, ίσχυσε στην περίπτωση των ε, ανακοινώσεων αλλά όχι στην περίπτωση του πυρηνικού. Εμείς ε, θελήσαμε να, να κουτσουρέψουμε τον προϋπολογισμό, να μιλήσουμε, να, να αφιερώσουμε αυτά τα ποσά για την καταπολέμηση των ε, επιπτώσεων της πυρηνικής ενέργειας. Εσείς μας λέτε ότι και μάθαμε από την Φουκουσίμα ότι δεν είχαμε πολλούς αρμόδιους στον τομέα, ανθρώπους ικανούς και εκπαιδευμένους για την εμπειρογνώμονες για την αντιμετώπιση μιας πυρηνικής κρίσης, για να αξιολογήσουν τη δόση, να δούνε τι γίνεται. Σχετικά τώρα με το κλείσιμο. Καμία, κα, κα, κανένα πυρηνικό εργοστάσιο δεν έκλεισε. Ως Γαλλίδα, μόνο το Μπρενελής ε, αρχίζει να διαλύει ε, το, τον αντιδραστήρα του από, τις 50, από τα 54 πυρηνικά εργοστάσια τα οποία έχουμε. Η Ευρώπη θα έπρεπε να είναι πρωτοπορία, ούτω ώστε το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων να ε, αποτελέσει παράδειγμα για το μέλλον, για το κόστος της έρευνας, μα είναι η διάφορη λειτουργία που πρέπει να το... Οι διάφοροι προμηθευτές είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να ασχοληθούν και με την έρευνα και με τη διαχείριση των αποβλήτων, όχι ο καταναλωτής. Και επίσης το θέμα των ε, ε, μηχανών και εργα... διαπίστωσης ε, της ραδιενέργειας. Σε ένα εργοστάσιο που κατασκεύαζε τέτοιου είδους μηχανήματα δημιουργήθηκε ένα νέφος και δεν ξέραμε από ποια ήταν η πηγή της μόλυνσης και γιατί, γιατί δεν είχαμε εμείς ε, τα, τα, απαραίτητα μέτρα, τα απαραίτητα όργανα για τη μέτρηση. Ζητούμε για το ΙΤΕΡ ενίσχυση από την Κομισιόν. Το ΙΤΕΡ πρέπει να χρηματοδοτηθεί εκτός των κοινοτικών προγραμμάτων, διότι πρόκειται εδώ για μια ομάδα ε, συμφερόντων που δεν έχει δουλειά. Με την Ένωση. Ο κύριος Πρόντι, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεύμα εργασίας που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες με τον διευθυντή του ΚΚΕΡ για το θέμα του κλεισίματος των πυρηνικών εργοστασίων. Μία εκτίμηση μας λέει ότι χρειάζονται 500 δισεκατομμύρια ευρώ για το κλείσιμο των πυρηνικών εργοστασίων στην Ευρώπη και χρεια... πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να το λάβουμε ιδιαίτερα στα σοβαρά και πιο συγκεκριμένα γιατί εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε μία κληρονομιά αυτού του στυλ στις μελλοντικέ γενιές και θα πρέπει υπεύθυνα να λάβουμε υπόψη μας την ανάγκη έρευνας για το πώς ε, θα τακτοποιήσουμε τα απόβλητα, πώς θα συσκευάσουμε αυτά τα απόβλητα, διότι για να μην έχουμε ε, παρά έναν ελάχιστο κίνδυνο ρήπανσης. Πρέπει λοιπόν σε αυτόν τον τομέα να προωθήσουμε όσο το δυνατόν την έρευνα και την εφευρετικότητα και τις ε, τεχνολογίες, τις ε, απαραίτητες τεχνολογίες για να ελαχιστοποιήσουμε το, τις ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις για πολλά χρόνια. Χωρίς μικρόφωνο πρόεδρος. Ο κύριος έλεγχ. Καταρχήν θα ήθελα την πρόταση Σκίνερ, να, να συγχαρώ για αυτή την πρόταση. Τον προβληματισμό τον θέτει στο σωστό πλαίσιο όσον αφορά την Ευρατόμ. Χωρίς, ας το πω έτσι, με ιδεολειπτικό τρόπο να προδικάζει οτιδήποτε. Για την ομάδα του ΕΛΚ θέλω να αποσαφηνίσω κάτι. Ότι την πυρηνική ενέργεια και την πυρηνική τεχνολογία την θεωρούμε μια αναγκαία τεχνολογία γέφυρας, γεφυροποίησης Απλά μπορώ να πω ότι σήμερα στην εκλογική μου περιφέρεια στη Γερμανία εδώ και 1,5 χρόνο έχουν αυξηθεί κατά πολύ σημαντικό ποσοστό οι τιμέ τη ηλεκτρική ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματο. Θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσουν όλα αυτά να αντισταθμιστούν με άλλε πηγέ ενέργεια, π.χ. ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια αρνούμε να δω το, τη σύμβαση Ευρατών και την πυρηνική τεχνολογία με μια ημερομηνία λήξης. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Είναι κοινικό όμως ότι αφενός οι πράσινοι απαιτούν τον τερματισμό της πυρηνικής ενέργειας, από την άλλη πλευρά όμως το θέμα της αποθήκευσης πυρηνικού υλικού και για την έρευνα και στα κράτη-μέλη το τροχοπεδούν και δεν το αφήνουν να προχωρήσει θα πρέπει τελικά να δούμε τι θα γίνει σε σχέση με τη συνθήκη Ευρατόμ και πώς θα προχωρήσουμε. Και για το ΙΤΕΡ, δύο λόγια. Το έχω αναφέρει επανειλημμένα στο παρελθόν. Εδώ έτσι χαλαρά λέγεται ότι χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για το ΙΤΕΡ. Όμως πρέπει κάπως πιο διαφοροποιημένα να δούμε το πράγμα. Όποιος δει τη συνθήκη της ε, σύμβαση ΙΤΕΡ, τη διεθνή αυτή συμφωνία, θα πρέπει να δει διαφοροποιημένα το θέμα. Ότι καταλήγει με ένα πλαίσιο συμφωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει απλά ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι διασφαλίσεις που καθορίζονται από αυτή τη συνθήκη θα πρέπει να υπάρξει χρηματοοικονομική αντιστάθμιση. Πολιτικά δηλαδή βρισκόμαστε σε μια φαιά ζώνη, σε ένα άγνωστο πεδίο αυτή τη στιγμή για τη χρηματοδότηση του 2020 θα ήταν αυταπάτη να νομίζει κανείς ότι το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται, ότι μπορεί δηλαδή να πάψει να υφίσταται. Θα ήμουν, κάτι, θα ήμουν απόλυτα εναντίον του αυτή την ε, κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει η κάλυψη αυτών των ε, χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σοντή. Δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Σοντή. για το ΙΤΕΡ. Να συγχαρώ τον εισηγητή και για τη θέληση, τη συμβιβαστική θέλωση που επιδεικνύει. Εγώ για την πρόταση να περάσει δηλαδή μέσω του Σεωρατώμα δεν συγχαίρω την Κομισιόν για αυτή την πρόταση να βγούμε, δηλαδή από τον κοινοτικό προπολογισμό, όταν η Κομισιόν κάθε φορά μας κάνει ένα κεφάλι καζάνι στις Ολομέλειες, μιλώντας για κοινοτικό κεκτημένο, κοινωνικό κεκτημένο, κοινωνικό κεκτημένο. Μα εδώ πρόκειται για ένα παγκόσμιο σχέδιο. Σας παρακαλώ, τι εικόνα θα δώσουμε άμα δεν είμαστε ικανοί να βρούμε 2-3 εκατομμύρια ευρώ που πρόκειται περί ε, ε, για κάτι το ιδιοφιές. Ε, ιδιοφιές όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά για την ανθρωπότητα. Δηλαδή πραγματικά η αδεξιότητα της Κομισιόν εδώ είναι ασύλληπτη. Εμείς Εγώ θέλω να συγχαρώ το ΚΚΡ το οποίο ε, επιτελεί εξαιρετικό έργο, αξιοποιεί ιδιαίτερα τη χρηματοδότηση αξιοποιεί τη χρηματοδότηση πολύ σωστά. Εμείς όμως ε, στα δύο χρόνια εδώ δίνουμε, δώσαμε στο παρελθόν μία παράταση δύο ετών. Δεν ξέρω εσείς όμως πώς μπορείτε να βρείτε μια καινούργια πρόταση για να έχουμε μία συνεκτικότητα στη διάρκεια, να έχουμε άλλα δύο χρόνια μετά. Θα ήθελα η Κομισιόν να δεχθεί τις τροπολογίες για τις οποίες ε, θα έχουμε ε, μεγάλη υποστήριξη Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει μία κοινοβουλευτική διάσταση. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι ήρθε πια η ώρα η συνθήκη ορατών να ενταχθεί υπό την ε, υπό τη συναπόφαση και η Κομισιόν να συμφωνήσει μια φορά μαζί μας για να δεχθεί όλες τις προτάσεις οι οποίες θα έχουν μια τέτοια διάσταση. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη για, τους, για τις παρεμβάσεις τους. Ο κύριος Κίνερ έχει κάνει μια πολύ ισόρροπη πρόταση. Πέντε βασικά σημεία οι τροπολογίε προσπαθούν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογή ή τον στόχο του, της του προγράμματος. Εμείς δεν τονίζουμε τόσο πολύ την πυρηνική τεχνολογία. Θέλουμε να παραμείνουμε στον πολιτικό συμβιβασμό που υπάρχει ήδη. Στο τελευταίο κομμάτι της Ευρατόμ ε, ακούστηκαν και τα stress test στην παρόδο. Ε, θα ήταν χρήσιμο σημείο, όντω. Ε, Αναφέρατε επίση και την κατάρτιση και την ασφάλεια, κύριε Σκίνερ. Σωστό, καλώ το κάνατε. Είναι σημαντικό θέμα. Επίση. of course, there is research and development as a Η πάυση λειτουργία ήταν πολύ σημαντική. Οι βιομηχανικές ε, δραστηριότητε βεβαίω είναι λίγο διαφορετικές. Εδώ ξεπερνούμε λίγο την έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω το αναφέρατε, και, το αναφέρατε μερικοί από εσά στην διαφάνεια, ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλέκεται ενεργά και στενά. Ε, αυτό το θέμα είναι θέμα θεσμικό, έχουμε μια συνθήκη, σε αυτή βασιζόμαστε, σε από αυτήν εξαρτώμεθα και εμείς ως Κομισιόν Βεβαίω θα, θα συνεχίσουμε να προσκαλούμε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει, οπότε να είσαστε σίγουροι ότι υπάρχει κατανόηση αμοιβαία και λαμβάνουμε υπόψη τα σχόλιά σας. Για την ε, μείωση τώρα, ε, τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογή και του προπολογισμού. Αυτό ας το κρατήσουμε. Θέλουμε να είμαστε και σε συνέφεια με τους βασικούς στόχους του ορίζοντα 2020 και κυρίως στους τρεις βασικούς πυλώνες. Ε, αριστεία, ε, αρχηγία, ηγεσία και ε, κοινωνικές προκλήσεις. Θέλουμε λοιπόν και το κομμάτι της, Euro, της που αφορά σε αυτό να αντικατοπτρίζει ακριβώς τον, τους τρεις αυτούς πυλώνες του ορίζοντα. Επίσης, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες που ξεκινούν από, τις, από κάποια οριζόντια σημεία στον ορίζοντα, α πούμε διεθνή συνεργασία, θέματα φύλου, μικρομεσαίες επιχειρήσει κλπ. Α προσπαθήσουμε να είμαστε συνεκτικοί σε αυτά τα δύο. Μετά, ίτερ. Προφανώ, ε, το γνωρίζετε ποια είναι η θέση τη Κομισιόν. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εκπέσει του MFF. Έχουμε προτείνει ένα επιπλέον πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη και υπάρχει και αρκετή επιχειρηματολογία υπέρ αυτού. έχουμε αυτό το θέμα τώρα της εφταετίας ε, έναντι της πενταετίας. Τεχνικά, λόγω της ε, συνθήκης, έχουμε 5 συν 2. Αλλά έχουμε και το earmarking, ε, το συγκεκριμένο, τη στοχοθέτηση των κονδυλίων για, για τα 7 χρόνια. Οπότε έχουμε έτσι μια καλή άποψη για αυτά τα δύο εναπομείναντα έτη. Ευχαριστώ όχι, να απαντήσω λίγο σε αυτό που είπε ο Κομισιόν. Το νομικό ερώτημα, σε ποιο βαθμό, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση για, την, για το ίτερ, λόγω των, λόγω το, αν δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το ίτερ από, την, από την χρηματοδότηση της Κομισιόν, πάει πίσω στην χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Ε, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα this, this was really good question. Καλή ερώτηση κάνατε, κύριε Έλλερ. Skinner, you want to sum up? Κύριε Σκίνερ. Του κάνατε πολύ καλή τρίπλα, κύριε Έλλερ, του εκπροσώπου της Κομισιόν. Λοιπόν, ε, θέλουμε όντως να... Ε, αυτό που λέει η Κομισιόν μάλλον δεν ε, είναι έτσι λάθος. Όντως ε, πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα και πρέπει να προχωρήσουμε. Εντάξει, ίσως σε κάποια σημεία παρακλίνουμε λίγο από αυτό που είχα προτείνει εγώ, αλλά νομίζω ότι θα ξεκολουθήσουμε να είμαστε επιτυχείς ε, για τα προγράμματα που έχουμε προτείνει. Τώρα, για κάποια από τα σημεία που ακούστηκαν ε, ε, μιλήσαμε για την συνθήκη τη Ευρατόμ, για την πάυση της λειτουργίας και για τις ε, θέσει εργασίας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να καταρτήσουμε κάποιους, όχι μόνο πυρηνικού επιστήμονες, αλλά να βοηθήσουμε και την, ε, και την πάυση της λειτουργίας. Δεν, δεν μπορώ να συμφωνήσω να φύγει η κρατική χρηματοδότηση. Από την αρχή ε, παρεμβαίνει, υπάρχει κρατική χρηματοδότηση. Αυτό που λέμε είναι ότι ουσιαστικά σκοτώστε την πυρηνική βιομηχανία. Δυστυχώ δεν μπορώ να συμφωνήσω εγώ με αυτό. Το κόστο τη ενέργεια που είπε ο κύριο Έλερ. δεν μπορούμε να προσποιούμεθα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο τι συμβαίνει. Ε, Βιτόριο, χάρηκα με αυτό που είπες, θα το συμπεριλάβω για τον επικεφαλής ε, του, της συγκεκριμένης επιτροπής που ήρθε και σου μίλησε για την σημασία των κονδυλίων που θα αποδοθούν. Ε. Εδώ μιλούμε για το ότι πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Πρέπει να δείξουμε αποτελέσματα και πρέπει αυτά τα αποτελέσματα να έχουν και προσθέμενη αξία. Κρίστιαν, ε, έχεις δίκιο. Ε, μίλησες για τις, ε, ε για τις ε, εκλογικέ μας περιφέρειες. Είπες ότι μέσα σε 16 μήνες αυξήθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού 50%. Ε, προφανώς θέλουμε και εμείς να υπάρχει όφελος για τους πολίτες. Βεβαίως πρέπει να ξέρουμε και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα αλλά ας τονίσουμε περισσότερο το ότι υπάρχει και ένδια ενέργειας Στι χώρες μας και εμείς ε, στη χώρα μου εισάγουμε την περισσότερη μα ενέργεια και προφανώς ε, αυτό ε, εκτινάσει και τις τιμέ. Γνωρίζω λοιπόν το τι γίνεται και ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες εκλογικέ περιφέρειες που πιστεύουν το ίδιο. Κύριο Ντία, συμφωνώ με αυτό που λέτε για το ότι υπάρχει έλλειψη συνοχής για το θέμα του προπολογισμού. Σε ένα βαθμό έχω πιέσει όσο μπορούσα, αλλά όπως έχουμε πει και σε άλλες ε, επιτροπές, το έχουμε ξανασυζητήσει, η κυρία Χέρτσοκ δεν είναι εδώ, είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Έχει υποσχεθεί ότι θα ε, προσπαθεί να πιέσει έτσι ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση, αλλά η πίεση βεβαίω βρίσκεται στο Συμβούλιο που πρέπει να βρει τα κονδύλια. Οπότε νομίζω ότι εδώ έχουμε ακόμα κάποιο περιθώριο ε, πίεση. Ευχαριστώ κύριε Σκίνερ. Τελευταίο σημείο. Η αιτήση. Για πέντε λεπτά θα λάβει τον λόγο εισηγητής ο κύριος Κρόισμαν. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σας ευχαριστώ. Προσπάθησα στις προτάσεις που υπέβαλα για τους νόμιμους ελέγχους των ετήσιων λογαριασμών να πετύχω την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών, την ενδυνάμωση των επενδυτών, δηλαδή των ιδιοκτητών και την ανεξαρτησία των ε, ελεγκτών, των οικονομικών ελεγκτών. Θέλω να πω, εκινώντας από αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, <clears throat> εκινούσε από μια χρηματοοικονομική κρίση και ήθελε να αναλάβει την προσπάθεια το λιγοπόλιο των τεσσάρων μεγάλων οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης ε, να το ε, σπάσει. Και καταλήγουμε στην πρώτη πρόταση αμέσως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή υποχρεωτική ανακύκλωση. Και έκανα πολλές συζητήσεις και μετά από έξι χρόνια <clears throat> ο στόχος που θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αμφιβάλλω αν μπορεί να επιτευχθεί. Πρέπει να το δείτε αυτό. Χρειάζεται τρία-τέσσερα χρόνια ο οικονομικός ελεγκτής για να μπορέσει να αναλύσει μια πανεθνική, μια πολυεθνική επιχείρηση και να καταλήξει στο ότι έχει γίνει μια σωστή ανάλυση και μετά από μια υποχρεωτική ανακύκλωση έξι ετών θα χάναμε το στόχο και θα υπήρχε ο κίνδυνος υπό όρους και προϋποθέσεις αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μπορεί να επιτευχθεί. Το δεύτερο είναι ότι με μια υποχρεωτική ανακύκλωση θα μπορούσε να καταλήξει κανείς στο ότι από τους τέσσερις ε, μεγάλους οίκους θα μπορούσαν να 5, 6, 7. Δεν νομίζω ότι αν χάσει την εντολή της ε, ένας μεγάλος οίκος μετά θα, έχουμε κάποια ε, ανατροπή των πραγμάτων και μάλιστα εις βάρος του καθεστώτος των μικρομεσαίων. Θέλω να υπάρξει κινητοποίηση των πραγμάτων με την ανεξαρτησία των οικονομικών ελεγκτών, με μια υποχρεωτική υποβολή προτάσεων και προσφορών. Θα πρέπει μετά από 7 χρόνια να υποβάλλονται προσφορές και αν μετά στις επιχειρήσεις από πλευράς των ίδιων οίκων θα πρέπει να παραμείνουν στους ίδιους οίκους, θα πρέπει στους μεριδιούχους να τεκμηριώσουν πολύ καλά αυτή την πρόθεση και τότε θα υπάρχει δυνατότητα να πει κάποιος ότι θέλω να παραμείνω στον ελεγκτικό αυτό οίκο ή όχι. Μετά όμως από 14 χρόνια πιστεύω ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια αλλαγή οικονομικών ελεγκτών. Γι' αυτό η πρόταση είναι μία φορά μετά από επταετή περίοδο να μπορεί να παρατείνεται αυτή η περίοδος ώστε μετά από δύο φορές επταετή περίοδος, μετά από 14 χρόνια να μπορεί να αλλάξει ο οικονομικός ελεγκτής. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα ανεξαρτησίας και στους οικονομικούς ελεγκτές. Και γι' αυτό ακολουθεί αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια ε, πρόταση ε, τροπολογίας θα υποβάλουμε εμείς πρόταση για τριετή περίοδο. Η προστασία των επενδυτών ήταν κάτι το οποίο θέλαμε να πετύχουμε και όποιος θέλει να πετύχει αυτόν τον στόχο, οπωσδήποτε χωρίς αμφιβολία, το, το Συμβούλιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει αυτή την πτυχή. Γι' αυτό μετά από τρία χρόνια το ελεγκτικό έργο των οικονομικών ελεκτών σε τακτά διαστήματα από την Ελεκτική Επιτροπή ε, θα πρέπει να ε, εποκτεύεται, να, να, ελέγχεται και σε περίπτωση ακραία θα μπορούσε να υπάρξει ανακύκλωση ε, ελεγκτικών αρχών, ιδιωτικών τέτοιων υπηρεσιών πριν από την τριετή περίοδο. Αυτό μπορεί να γίνει από την Εποπτική ε, Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται μια, ένα διαφανές πλαίσιο εποπτείας. Πιστεύω ότι από πλευράς της Επιτροπής ε, θα πρέπει να διασφαλίζονται όλα αυτά και μέσω μιας ε, δημόσιας υποβολής προτάσεων πρέπει να διασφαλίζεται η υλοποίηση αυτών των στόχων. Θα επιτρέπεται ο καλύτερος ανταγωνισμός και η βέλτιστη επιλογή. Και θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα οποία δεν συναποτελούν ε, μέρος των ε, ελεκτικών δραστηριοτήτων να μην εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό με οδηγεί αμέσω ε, στο θέμα της παροχής υπηρεσιών. Τρεις κατηγορίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θετικά για τους ελέγχους, αρνητικά για τους ελέγχους και μια ενδιάμεση κατηγορία όπου θα μπορεί να υπάρχει η εποπτική αρχή που θα διασφαλίζει αν κάτι είναι θετικό ή αρνητικό. Θέλουμε να υπάρχει μείωση της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και γι' αυτό προτείνουμε δύο κατηγορίες να υπάρχουν και όχι τρεις. Δηλαδή, εξέταση των υπηρεσιών που θα εγκρίνονται και θα παρέχονται και αρνητικές εις βάρος των υπηρεσιών ε, υπηρεσίες. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μικρότερη γραφειοκρατική επιβάρηση. Οι ελεγκτικές εταιρείες θα ξέρουν τι μπορούν να προτείνουν και τι μπορούν να ελέγξουν ως παροχή υπηρεσίας και πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά ώστε να μπορεί να συντάσσεται, να δίνεται η καλύτερη εντολή ελέγχου. Είναι αυτονόητο ότι σε αυτή την πρόταση υπάρχει και το θέμα του ορίου. Αυτό είναι πολλές φορές προβληματικό, οδηγεί σε γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Δύο λόγια για τον κανονισμό, Πρόεδρε, που πρέπει και αυτό να καλύψω ως θέμα, το θέμα του κανονισμού. Και εκεί έχουμε μια συμμετοχή στο κεφάλαιο που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φυσικά αν 100% κεφαλαιακή απέτηση ε, προϋποτίθεται, τότε μπορεί αυτό να είναι επιβάρυνση. Γι' αυτό εγώ θα προτείνω μέχρι 49% κεφαλαιακή συμμετοχή. Ο καθορισμός, η απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των οικονομικών ελεγκτών και γι' αυτό 100% των ε, δικαιωμάτων ψήφου θα πρέπει να διασφαλίζονται σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κρόιτσμαν. Ο κύριος Σοντή. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε συγγνώμη για τον συνάδελφο, για τον, τον κύριο Φράνκρουστ, ο οποίος απουσιάζει, όπως επίσης και η συντονίστρια. Και επειδή όπως είδατε δεν υπάρχει κανένας, με στείλανε επί... Με στείλανε για να πω εγώ τη γνώμη της ομάδας. Βέβαια υπάρχει εδώ ένα σύμβατο, διότι και εγώ είμαι ελεγκτής. Λοιπόν, Πρέπει ε, να, να, προσέξει ο εισηγητής ότι ο έλεγχος, το audit λειτουργεί κανονικά, ο ανταγωνισμός λειτουργεί κανονικά. Ο εμείς ε, θα υποστηρίξουμε μεγάλο βαθμό των προτάσεων του εισηγητή. Θα καταθέσουμε τις ε, τροπολογίες που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες για αυτό το ντοσιέ. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις επί της για τις υπηρεσίες του, μη ελέγχου θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε από τις υπηρεσίες ελέγχου και επίσης να δούμε το θέμα της εποπτείας των αρχών που ελέγχουν τους ελεγκτές. Ίσως να φαίνεται αυτό ιδιαίτερα πολύπλοκο, αλλά για να συνεννοηθούμε κάθε μέρα τι γίνεται. Έχουμε εμείς υπερεθνικές επιχειρήσεις που έχουν έναν ελεγκτή. Δηλαδή οι επιχειρήσεις ε, audit ελέγχου έχουν υπερεθνικές αρμοδιότητες. Ποιος θα ελέγξει τον, τον ελεγκτή. Και υπάρχει κάτι στην πρόταση που δεν αντιμετωπίζεται σωστά, είναι το ποιος εποπτεύει τις υπερεθνικές ελεγκτικές εταιρείες είναι το ίδιο με τη συζήτηση που είχαμε δηλαδή για την Τραπεζική Ένωση. Εμείς ε, μιλάμε να έχουμε μία ενιαία εποπτεία των ε, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και βλέπουμε την Κομισιόν να είναι αρκετά συγκρατημένη λέγοντας ότι εδώ παίζει ο συντονισμός. Ή εμείς θεωρούμε ότι η χρηματοπιστωτική αρχή είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ελέγχει όλους αυτούς τους ελεγκτές ε, που ελέγχουν υπό την Ευρωπαϊκή Αρχή τις ελεγκτικές αρχές. Λοιπόν, πρέπει να δούμε τι γίνεται για τον υπερεθνικό έλεγχο εποπτείας των ελεγκτών για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε και την ποιότητα εργασίας των ελεγκτών. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή, τον κύριο Κρότσμαν, για όλε τι ε, προσπάθειες που έκανε να υποστηρίξει αυτή τη μεταρρύθμιση του τομέα του λογιστικού ελέγχου, ώστε να επιτύχει του στόχου του. Ο κύριος ε, Κρόιτσμαν και η έκθεση του τονίζουν ότι το status quo δεν είναι επιλογή και δείχνει η έκθεση ότι οι στόχοι της μεταρρύθμισης που όντω θα βελτιώσουν την ε, ποιότητα των λογιστικών ελεγχών στην Ένωση και θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά και την οικονομική σταθερότητα, είναι ένα κοινό τόπο. Ε, μια που είναι περιορισμένο ο χρόνο μου, εμεί ε, δεν θα σχολιάσουμε το κάθε μικρό σημείο που υπάρχει στην, στο σχέδιο έκθεση. αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ στα βασικά σημεία, στα σημεία κλειδιά που έθεσε και ο κύριο Κρόιτσμαν και ο κύριο Οντί. Πρώτον, Όπω τονίζει πάντα η Κομισιόν και τονίζεται και στην έκθεση Κρόιτσμαν, η ανεξαρτησία των ελεκτών είναι σημείο ουσία για την ποιότητα του λογιστικού ελέγχου. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι ε, αρχή της, γι' αυτό θεωρούμε ότι η αρχή της υποχρεωτικής ε, ε, περιτροπής είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε απειλή ή κίνδυνο και να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία των ελεγκτών. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε ε, την μέγιστη δυνατή δέσμευση για τους ελεγκτές. Οπότε η Κομισιόν καλωσορίζει την πρόθεση που έχει ο εισηγητής ε, να υποβάλει κάποια συμβαστική πρόταση ως προς αυτό. Επίσης, σημειώνουμε την ε, πρόταση που γίνεται μέσα στο σχέδιο γνωμοδότησης ότι η διάρκεια μιας δέσμευσης ε, λογιστικού ελέγχου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 7 χρόνια που θα μπορεί να ανανεώνεται άπαξ. Κατά συνέπεια η υποχρεωτική περιτροπή θα, γίνεται, θα είναι για 14 χρόνια. Το σημειώνουμε αυτό ως ένα στοιχείο συμβιβασμού Βεβαίως ε, στη φάση αυτή δεν είναι δυνατό να πάρει θέση η Κομισιόν επ' αυτού, αλλά το σημειώνουμε. Επίσης πρέπει να τονίσω το ότι στην αρχική πρόταση της ε, Κομισιόν ο κοινό ε, λογιστικός έλεγχος ε, προτινόταν με κάποια κίνητρα και στην αρχική πρόταση Κομισιόν η αρχική δέσμευση ήταν 6 χρόνια για το λογιστικό έλεγχο. παρόλα αυτά για τους κοινού λογιστικούς ελέγχους αυτά τα 6 χρόνια γίνονταν 9 χρόνια το ανώτερο. Οπότε εμείς λυπούμεθα λίγο για το ότι ε, η πρόταση της γνωμοδότησης του κυρίου Κρόιτσμαν δεν δίνει κάποιο κίνητρο για, τα, για τους κοινούς λογιστικούς ελέγχους. Σχόλια του κύριου Κρότσμαν χωρίς μικρόφωνο. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα. Ε, ε, η Κομισιόν καλωσορίζει το γεγονό ότι ε, η γνωμοδότηση θέλει να ενισχύσει την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή συνεργασία και αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Η Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου πρέπει να έχει τι αρμοδιότητε που τι αρμόζουν για να μπορεί να, κάνετε, να εκτελεί τα καθήκοντά τη. Τώρα, για, ε, για τι υπηρεσίε μη λογιστικού ελέγχου. Η Κομισιόν κατανοεί ότι αυτέ οι υπηρεσίε που απαιτούνται ε, που απαιτούνται να γίνουν από τους ελεκτές δυνάμει του εθνικού δικαίου θα πρέπει να επιτρέπονται. Απ' την άλλη, η η, η προσφορά κάποιων υπηρεσιών, όπως οι φορολογικές συμβουλές ας πούμε, και η ε, συμμόρφωση με τις ε, φορολογικές απαιτήσει που ξεπερνούν τα όσα προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, αποτελεί απειλή για την ανεξαρτησία των ελεκτών. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών ενισχύει τις ε, δυνατότητες αυτορύθμισης ή βάζει τον τον ελεγκτή να πρέπει να υπερασπιστεί τις εταιρείε που ελέγχει. Που ουσιαστικά σημαίνει ότι περιορίζει την ανεξαρτησία του λογιστικού του ελέγχου. Για να ενισχύσουμε την επικοινωνία, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τις εκθέσεις των ε, ελεγκτών προς το κοινό. Η Κομισιόν κατανοεί και εκτιμά ότι αυτό αυτό είναι ένα από του στόχου που θέλει να επιτύχει ο εισηγητή. Οι εκθέσει του λογιστικού ελέγχου θα πρέπει να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίε στο κοινό, ώστε να μπορούν να πληρούν τον σκοπό του. Επομένω, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν παρέχουμε έξτρα πληροφορίες μόνο στις εσωτερικές εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου. Μόνο η Επιτροπή Ελέγχου θέλει ε, περισσότερε πληροφορίε και κάποιε πληροφορίε από αυτέ τι θέλει και το κοινό. Κύριε Κρότσμαν, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον για αυτό το θέμα της υποχρεωτικής ε, ανακύκλωσης ε, ε, να συζητήσουμε. Το σκέφτηκα, προβληματίστηκα για το joint audit. Στην Γαλλία είναι, έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το οποίο στο τέλος αναφέρατε, δηλαδή από τους εξωτερικούς ελέγχους σε σχέση με την πιστοποίηση να εξαιρεθούν κάποια πράγματα, σε σχέση με την περίπτωση Κιέρχ, στην Γερμανία αναφέρθηκε, δηλώθηκε επίσημα ότι είχε λέει προβλήματα η εταιρεία Kiers. Στη συνέχεια υπέβαλε αίτημα πτώχευσης ε, η εταιρεία αυτή. Αν δει κανεί ε, τώρα σε σχέση με το, ε, την ε, διακύβευση της επιχείρησης, δηλαδή αν διαπιστωνόταν, αν μπορούσε να διαπιστωθεί ότι βρισκόταν μπροστά στην πτώχευση η εταιρεία αυτή, Προτείνω να μην το κάνουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο γιατί μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα. Τα υπόλοιπα μπορούν να λειτουργήσουν. Αν υπάρξουν κάποια σφάλματα, για παράδειγμα, στο, στους υπολογισμούς, δεν πρέπει να δημιουργούνται λανθασμένες ε, προσδοκίες από μια τέτοια πιστοποίηση. Γι' αυτό αφαίρεσα από την πιστοποίηση αυτά τα θέματα και τα έθεσα στο θέμα, στο πλαίσιο εκείνο που έχουν υποχρέωση οι ελεγκτές με κάθε σθένος ε, να ελέγχουν. Κατά τα άλλα θα παραμείνουμε σε συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το θέμα των εταιριών ελέγχων να μπορούν να ελέγχονται εθνικά αυτές οι δράσεις στην Γερμανία με την αρχή εποπτείας των χρηματοοικονομικών αυτών ε, ε, οργάνων. Όταν υπάρχουν κάποια προβλήματα μπορεί να ληφθεί η απόφαση αλλαγής οργάνου. Φυσικά δρούν παγκόσμια τέτοιου είδου επιχειρήσει. Υπάρχει όμω και η εθνική εποπτεία. Είναι όμω το τέλο τέλο υπεύθυνοι για αυτέ τι ε, πιστοποιήσει, για αυτά τα στοιχεία τα οποία ε, πιστοποιούν στην Γαλλία ή στην Ιταλία όπου εκδίδονται. Γι' αυτό αυτό πρέπει να είναι αρκετή αφορμή για τις ε, κρατικές αρχές αυτών των κρατών, αν δεν υλοποιούνται επαρκώς ε, οι προϋποθέσεις ε, των ελέγχων, να αφαιρείται η εντολή τους. Κάθε τρία χρόνια είχα ζητήσει να γίνεται αυτό. Δεν το εμπεριείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Πρέπει να υπάρχει αυστηροποίηση λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο και πρέπει να σκεφτούμε ποιος θα επιβάλλει κυρώσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Θέλω να κάνω δύο ανακοινώσεις. Πρώτον, αύριο στις 10 το πρωί θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με ψηφοφορία. Δεύτερη ανακοίνωση. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για αυτή την έκθεση του κυρίου Κρόσμαν θα είναι η 16 Οκτωβρίου 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.